Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ρέντινγκ, αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ε, που ασχολείται κυρίως με θέματα ε, δικαιωμάτων ε, και πολιτών. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, κάποια μέτρα, κάποια κοινά μέτρα με την ε, κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ. Θα... Έχουμε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας σε σχέση με τον δομημένο διάλογο που γίνεται κάθε χρόνο ανάμεσα στις επιτροπές και τους αρμόδιους επιτρόπους σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και τις προτεραιότητες για τις ερχόμενες χρονιές. Έτσι έχει η Επιτροπή μας και την ευκαιρία να συζητήσει με την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ σχετικά με ε, τον χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών που υιοθέτησε η Κομισιόν στις 5 Μαρτίου. Ε, περιμένουμε να ακούσουμε τις πληροφορίες της κυρίας Ρέντινγκ. Θα έχουμε την ευκαιρία και να συζητήσουμε. Θα τις δώσω το λόγο Ορίζοντας, την Επίτροπο. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ladies. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, που δεν είναι πολλοί, αλλά πάντοτε, αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους άντρες στην Επιτροπή Γυναικών, αλλά αυτό τόσα χρόνια, 20 χρόνια το λέω. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους προσελκύσουμε. I great importance uh, to develop very good with... Θα ήθελα να αναπτύξουμε ιδιαίτερα καλές σχέσεις ε, εσείς και εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν κοινό αγώνα. Έχουμε συνεργαστεί καλά και στη Νέα Υόρκη στην υψηλού επίπεδου διάσκεψη των ΗΕ Εθνών για την κατάσταση των γυναικών. Ήσασταν και εσείς εκεί. Είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και με γυναίκες από όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πτυχή της δουλειάς μας. Θα θυμάστε, κυρία Πρόεδρε, το ετήσιο πρωινό μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και Επιτροπής Γυναικών ε, όπου ανέφερα τις προθέσεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια είχαμε και τις, τις ακροάσεις, ε, την ακρόασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν τόσο επικοδομητικοί. Από τότε όμως έχει περάσει πολύ καιρός και έχουμε κάνει και πολλά μαζί. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι προκλήσεις δεν είναι λιγότερες, αλλά περισσότερες. Γιατί τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας είναι αυτά που καθίστανται πιο ευάλωτα σε περιόδους κρίσεων και αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση με τα πολλά προβλήματα που πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε, όπως για παράδειγμα πλήρη ισότητα των φύλων στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, όχι μόνο στα χαρτιά. Και νομίζω ότι δεν, γίνεται, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλέον δικαιολογίε ε, για θύματα βίας, ε, ε, γυναίκες θύματα βίας, γυναίκες που ζουν στη φτώχεια, χάνουν τις δουλειές τους επειδή μένουν έγκυες ε, ή για άλλους πολλούς λόγους. Όσον αφορά τώρα το νομοθετικό πλαίσιο, η εφαρμογή και η ενίσχυση των νομικών δικαιωμάτων των γυναικών ε, είναι μία από τις πρώτες και απόλυτες προτεραιότητες μου. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες ε, που έχουμε ήδη όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της οδηγίας για τη γονεϊκή άδεια που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ευθύνη των ε, πατέρων ε, για ε, τα παιδιά τους. Επίσης έχουμε δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή που επεξεργαζόμαστε. Πρώτον, η προστασία των εγγύων γυναικών και δεύτερον, των αυτοαπασχολούμενων και των γυναικών Uh, των γυναικών ε, συνεταίρων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό ε, στο πλαίσιο της ε, βιωσιμότητας της κοινωνίας μας. Επίσης, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι προσφάτως είχαμε μία συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό τομέα και η ανάλυση, σύμφωνα με την ανάλυση μας είναι ότι όλοι οι κλάδοι στους οποίους υπάρχουν, ε, υπάρχει ισότητα των φύλων έχουν και μεγαλύτερα έσοδα. Αυτοί λοιπόν που δεν φοβούνται τις γυναίκες ε, τα πάνε καλύτερα. Και αυτό είναι κάτι που συχνά ξεχνούμε να τονίσουμε. Οπότε και οι δύο αυτές οδηγίες για τις ε, έγκυες γυναίκες και για τις ε, αυτοαπασχολούμενες εξασφαλίζουν υψηλότερο ποσοστό ε, απασχόλησης των γυναικών αλλά και μεγαλύτερη ισορροπία με, στο πλαίσιο της κοινωνίας, της, των χώρων εργασίας και έχουμε, και συμ... έχουμε σημαντικούς, σημαντικές εβδομάδες και μήνες μπροστά μας για τις οδηγίες αυτές και θα ήθελα να υποστηρίξω την κυρία Λούλιν και την κυρία Εστρέλα στις ε, ζωτικής σημασίας προσπάθειές τους ε, να συμφωνήσουμε το Συμβούλιο. Δεν θα είναι εύκολο. Τώρα, Όσον αφορά τώρα την επιτυχία για την οδηγία γονεϊκής άδεια, πρέπει να δούμε και άλλου είδους άδειε που μπορούν να υποστηρίξουν τη ισότητα των φύλων. Γνωρίζετε ότι η πατρική άδεια δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην ε, άδεια των εγγύων γυναικών, γιατί το θέμα είναι θέλουμε ή δεν θέλουμε. Θέλουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο αν θέλουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, μπορεί να πρέπει να μειώσουμε κάπως τους στόχους μας. Αλλά έχω κάθε πρόθεση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να συζητήσω ένα ευρύτερο θέμα. Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια πολιτική για να ενισχύσουμε τους... Ε, για να ενθαρρύνουμε τους πατέρες να λαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες για τα παιδιά τους. δεν θα είχα κάνει όλα αυτά, όσα, όλα αυτά που έκανα, να μεγαλώσω τρία αγόρια, να είμαι πολιτικός, δημοσιογράφος, αν ε, δεν ε, είχα δίπλα μου έναν πατέρα που ε, ασχολείται με τα παιδιά του. Είναι ο μόνος τρόπος για να, για να επιτύχουμε. Άκουσα τις ανησυχίες σας και ζήτησα και από τις υπηρεσίες μου να κάνουν μια εις μελέτη για το και τη σχέση κόστους και ωφέλους των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών που έχουμε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε απλώς επιθυμούμε κάτι. Πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας. Και σίγουρα θα είδατε ότι έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011. Όσον αφορά τώρα περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες, εγώ θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας ε, ιδέες. για να μπορέσουμε να έχουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν τομείς για τους οποίους θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, το θέμα των ποσοστώσεων. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση των μισθολογικών διαφορών. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι φορείς που ασχολούνται με την ισότητα πρέχουν τους πόρους, την ε, δύναμη και την ανεξαρτησία να κάνουν τη δουλειά τους. Χρειαζόμαστε αυτούς τους ε, φορείς ε, να διαδραματίσουν δηλαδή τον πλήρη ρόλο τους. Και γι' αυτό ακριβώ θα δρομολογήσω σχετική νομοθεσία για όλου αυτού του τομεί. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή τη ε, νομοθεσία, το έχω πει πολλέ φορέ και θα το επαναλάβω. Μηδενική ανοχή όσον αφορά την έλλειψη εφαρμογής ε, της, ε, του κεκτημένου που ήδη έχουμε στον τομέα αυτό. Και εγώ ευχαρίστως να ακούσω πληροφορίες από εσά και ιδέες. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθώ να το προωθήσω, διαπραγματεύομαι και συζητώ με τα κράτη-μέλη. Δεν έχω σκοπό να φτάσουμε στο δικαστήριο. Προτιμώ να λύνουμε τα προβλήματα πριν. Να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να συζητώ με τα κράτη-μέλη προκειμένου να τροποποιήσουν την, τις νομοθεσίες τους. Θα ήθελα επίση, επί τη ευκαιρία, να πω ορισμένα πράγματα για τη χάρτα δικαιωμάτων των γυναικών ε, που παρουσίασα στι 5 Μαρτίου από κοινού με τον πρόεδρο Μπαρόσο. Η χάρτα αυτή για τα δικαιώματα των γυναικών Είναι μια νέα κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποτέ στο παρελθόν ε, δεν υποσχέθηκαν ε, όλοι οι επίτροποι από κοινού το ζήτημα της ισότητας των φύλων να συμπεριληφθεί σε όλες τις εργασίες τους. Είναι λοιπόν μια πολιτική δέσμευση κάθε μέλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρουν σοβαρά το θέμα των γυναικών ε, στα χαρτοφυλάκια τους. Πρόκειται λοιπόν για μία δέσμευση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι πράγματι θα συμβεί αυτό. Είναι μία πολύ σημαντική πολιτική πρωτοβουλία και πολλές άλλες που πρέπει κατά, τους, κατά τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να ε, να, να ληφθούν υπόψη, όπως για παράδειγμα ανεξαρτησία οικονομική, ε, ίση αμοιβή για, ίσα, για, για για ίση εργασία, ισότητα των γυναικών, ε, ισότητα στο πλαίσιο των συνδικάτων. Είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να μεταφραστούν στην πράξη. Και πρόκειται για μια νέα στρατηγική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η νέα στρατηγική θα αφορά όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και έχει να κάνει και με τον οδικό χάρτη 2006-2010 για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Θα σας παρουσιάσω τη νέα στρατηγική το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, θα έχετε πολύ σταθερή βάση για τις εργασίες σας. Ελπίζω επίσης ε, σε συνεχή διάλογο μαζί σας ε, για, ε, στο πλαίσιο του αγώνα μας για την ισότητα των φύλων και χαιρετίζω τις εργασίες της, του Κοινοβουλίου μέσω της έκθεσης κυρίας Φιγκουρέιντο για τα θέματα αυτά είπατε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας τριμερής διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χρόνο για την αναθεώρηση των πολιτικών ε, ισότητας των φύλων. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ καλό παράδειγμα. Να πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο, τις δεσμεύσεις των ε, διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων. Γιατί εμείς όλοι εδώ στη συγκεκριμένη επιτροπή συμφωνούμε και οι κυβερνήσει συμφωνούν μαζί μας. Στην, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλοι κάνουν τη δουλειά τους ε, προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μας υποστηρίζουν. Κάθε φορά που υποβάλλουμε μία νέα πρόταση. Όσον αφορά τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα υπάρξει και ένα πλαίσιο αντιμετώπιση τη βία κατά των γυναικών. Είναι κάτι που ζήτησε το Συμβούλιο Συμπεράσματά του όσον αφορά την εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών από το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στις, 6, στις 8 ε, Μαρτίου. Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεύρει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Κυρία Πρόεδρε, είδα, παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πόστερ, τις αφήσει που έχετε. Νομίζω ότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε την ιδέα αυτή για να ευαισθητοποιήσουμε και όλα στον κόσμο γιατί 25% των γυναικών έχουν ε, υποστεί βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και 10% έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής βίας. 6.000 κορίτσια κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο υφίστανται ακροτηριασμό γενετικών οργάνων. Είναι ένα φρικτό έγκλημα που δεν μπορούμε να το δεχόμαστε άλλο. Επίση, ε, θα προτείνω ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων ε, χωρίς ε, να αποκλείεται ευρωπαϊκή εναρμόνιση σε ποινικό επίπεδο όσον αφορά το θέμα των, του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα διασυνοριακά. Μία ακόμη προτεραιότητα για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μέχρι το τέλος της θητείας επιτροπής αυτής είναι 10%. Ξέρετε ότι δεν αλλάζει πάρα πολύ και σε μερικές χώρες μάλιστα γίνεται χειρότερο το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να σας το πω, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι κάτι το απαράδεκτο και πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να το καταστήσουμε προτεραιότητά μας. Παρακαλώ λοιπόν να κάνουμε αυτό που είπαμε στις 5 Μαρτίου όταν αρχίσαμε την εκστρατεία μας. Αυτό όμως είναι μόνο μια αρχή. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια ενημερωτική εκστρατεία και μετά να σταματάμε τις προσπάθειές μας. Πρέπει να συνεχίζουμε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε εγώ πάντοτε ευχαρίστως να σας ακούσω τι ιδέε σα πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτού του κοινού στόχου και πώ μπορούμε να προοδεύσουμε στο πλαίσιο της ε, κοινοβουλευτικής θητείας αυτής και της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ ε, σημαντικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και για τη δέσμευση που δείχνετε σε θέματα ισότητας. Η Επιτροπή μας προσβλέπει στην καλή συνεργασία στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά. να δώσω το λόγο στους βουλευτές για να συζητήσουμε και θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Γιάννα Κουδάκη, που είναι η υπεύθυνη στην Επιτροπή μας για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Παρακαλώ, κυρία Γιάννα Κουδάκη. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι θα μιλήσω πρώτη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στη συνεδρίασή μας ε, και σας ευχαριστώ και για τη μεγάλη σημασία που δίνετε στην Επιτροπή μας. Έχετε δίκιο, περισσότερους άντρες, αλλά περισσότερο από περισσότερους άντρες θα ήθελα περισσότερες γυναίκες καταρχήν, διότι δεν εκπροσωπούμαστε πολύ καλά. Ε, αν σκεφτεί κανείς πόσοι από, πόσες από είναι παρούσες θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία αφορούν μια μεγαλύτερη ομάδα. Ε, αυτό έχει να κάνει και με τη συμμετοχή των ανδρών. Νομίζω ότι ε, συχνά η Επιτροπή μας επικεντρώνεται πολύ στενά σε κάποια θέματα τα οποία δεν αφορούν συχνά την ευρύτερη κοινωνία. Εγώ θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να δω περισσότερες γυναίκε στην Επιτροπή μας και μετά περισσότερους άντρε. Μου άρεσαν οι προτεραιότητες που αναφέρατε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βία, την ε, εμπορία ανθρώπων. και τον ε, ε, γενετικό ακροτηριασμό, τον ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων. Είναι θέματα που αφορούν όλες τις γυναίκες, αλλά ε, κάποια θέματα αφορούν και τους άντρες. Ε, η, βία και η εμπορία ανθρώπων. Θα πρέπει να, να μην σκεφτόμαστε στενά στα πλαίσια του δικού μας του κουτιού των γυναικείων θεμάτων. Όσον αφορά την ε, την ε, άδεια κοίησης, ε, αν τη συνδυάσουμε με την άδεια, τη γονική άδεια των ανδρών, αυτό θα υποβαθμίσει την γονική άδεια των ανδρών και αυτό δεν το θέλουμε. Ε, πάντως νομίζω ότι γενικά η Επιτροπή μας συμφωνεί στα θέματα αυτά. Να προχωρήσω. Όσον αφορά την νομοθεσία, είπατε ότι θέλετε περισσότερη νομοθεσία για να ενθαρρύνετε περισσότερες γυναίκες ε, στην απασχόληση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι το θέμα δεν είναι μόνο η νομοθεσία, είναι και οι ίδιες οι γυναίκες. Πολλές γυναίκες δεν θέλουν να εργαστούν και αν είναι αυτή η επιλογή τους, ας είναι. Αν επιλέγουν να μένουν στο σπίτι και να κάνουν πολύ καλή δουλειά στα πλαίσια της οικογένειας επειδή αυτό θέλουν, αυτό δεν είναι κακό. Νομίζω ότι είναι λάθος από εμά ως Επιτροπή Γυναικών να υποβαθμίσουμε τις γυναίκες, να υποτιμούμε τις γυναίκες αυτές και να μην ε, τους ε, αποδίδουμε το σεβασμό που χρειάζεται. Όσον αφορά το χάρτη ε, για τα δικαιώματα των γυναικών, ξέρω ότι η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται πολύ για το θέμα αυτό και πάλι όμως από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι ένα πρώτο βήμα της Επιτροπής ε, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το πρώτο βήμα προτού αρχίσουμε να ζητάμε πολλά πράγματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο χάρτη, που, ε, τα, οποία δεν στηρίζουν απαραίτητα όλοι. Είμαι λοιπόν αρκετά ικανοποιημένη με το χάρτη και το τελευταίο ε, θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Φαίνεται να υπάρχει ε, ε, διάσταση όσον αφορά την, ε, το νομικό καθεστώ. Είχαμε συζήτηση για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο και, το, ε, η Κομισιόν δεν φαίνεται να συμφωνούν. Θα ήθελα πολύ να το ξεκαθαρίσουν το θέμα αυτό πριν έρθουν σε εμά. Αλλά όταν ξεκαθαριστεί το θέμα τη. Ε, εντολής και όταν βρούμε τη σωστή νομική βάση πιστεύω ότι θα, πρέπει να, θα μπορεί να εφαρμόζεται όχι μόνο για τη βία αλλά και για ε, την ε, εμπορία ανθρώπων, τον ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων, τα παιδιά κλπ. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιανακουδάκη. Να σας θυμίσω ότι έχουμε χρόνο μέχρι τις 10 ε, που θα πρέπει να ε, αποχωρήσει η κυρία Ρέντινγκ. Να δώσω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Γκυμάη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προέδρε, είναι μεγάλη τιμή, τιμή μάλλον, να σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή μας. Αναφερθήκατε σε πολλά σημαντικά θεμάτα. Ένα τα σημαντικότατα ήταν η ίση Ήρθα από την Ορβηγία. Η νορβηγική κυβέρνηση ετοίμασε μελέτη για τα φύλλα και την αμοιβή και δεν σχετίζεται με την εμπειρία η αμοιβή και την παιδεία. Θα έπρεπε να πληρώνονται το ίδιο άντρε και γυναίκε όταν κάνουν την δουλειά και του απασχολεί ο ίδιο εργοδότη. Το θέμα τη αμοιβή τονίζει τι διαφορέ που υπάρχουν. Ο Βλαντιμίρ Σπίτλα, ο προκάτοχός, στήμασε ανακοίνωση. Και Έντιτ Μπάουερ, συνάδελφος και φίλη, ετοίμασε μια πολύ καλή έκθεση. Εάν ακολουθήσουμε τους ρυθμούς, 70 χρόνια θα καλυφθεί η διαφορά αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα πρέπει να βρούμε καλύτερη λύση. Δεύτερον, ποσοστό ισότητας όπως αποκαλείται. Ο κ. Μπαρόσο δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο τρεις γυναίκες επιτρόπους είχε. Η κοινωνία των πολιτών εκινήθη και τον Βούλιο εκινήθη και κάποιοι πρωθυπουργοί άλλαξαν άποψη. Και αυξήθηκε ο έθιμος των γυναικών. Εξακολουθεί να είναι δύσκολο και τον 21ο αιώνα να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση των γυναικών. Πρέπει να το θυμόμαστε. Αν η έκθεση ταραμπέλα υλοποιηθεί, να είναι ένας άντρας και μία γυναίκα επίτροπη στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 50-50, τότε θα υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη χάρτα. Η χάρτα Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Γυναικών ήταν στο μανιφέστο Συριστικού Κόμματο στην Προκλητική εκστρατεία. Έγινε μεγάλη συζήτηση εκτενή στο κόμμα μα και υποσχέθηκε στο SND ο κύριος Μπαρόσο ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό της χάρτας και δεσμεύτηκε. Και εγώ επιθυμούσα διακαώς να ακούσω εσάς αγαπητοί επίτροπε να πείτε αυτό που είπατε στην ακρόαση, ότι είναι η χάρτα του κυρίου Μπαρόσο. Αν την έχει στερνιστεί και πιστεύει ότι είναι δική του ιδέα, θα είμαι πολύ ικανοποιημένη. Θέλω πιο συγκεκριμένα πράγματα όμω. 8 Μαρτίου έγινε συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, απουσίασα δυστυχώ. Ο συνάδελφός παρουσίασε το θέμα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών είχα την τύχη να συναντήσω στη Νέα Υόρκη. Πριν παρουσιαστεί όμως το έγγραφο δεν υπήρξε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, ούτε με την κοινωνία των πολιτών. Αγαπητοί Επίτροπε, χρειαζόμαστε μελέτη για τη χάρτα. Ενδελεχή. και διαβούλευση για να μπορέσουμε να συναθρήσουμε νομοθεσία και διαθέσιμα μέσα και να σχετιστεί η χάρτα με τη στρατηγική για το 2020 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η στρατηγική τη Λισαβόνα ήταν πιο ευαίσθητη όσον αφορά τη διάσταση του φύλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Δεν περιέχεται εκεί. Δεν υπάρχει ευαισθησία όσον αφορά την ισότητα των φύλων που αφορά την οικονομία και την απασχόληση. Και η Ευρωπαϊκή Χάρτα η ισότητα των φύλων, από ό,τι καταλαβαίνω, ακολουθεί τον οδικό χάρτη. Γιατί Μάθαμε το 2001 ότι υπάρχει δικός χάρτης. Εμπεριέχει πέντε σημεία. Πέντε με έξι σημεία. Έπρεπε να ακολουθούν. Ο Βλάντιμιρ Σπίτλα ετοίμασε τον οδικό χάρτη ισότητα των οφείλων. Έγινε διαβούλευση. Αλλά θα θέλαμε αυτό να προωθηθεί μέσα της χάρτας. Έρευνα, ανάπτυξη και μετανάστευση που θέσει στόχους του 2020. Θέλουμε να τεθεί και ισότητα των φίλων σας στόχος και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. θέλουμε να γίνει διαβούλευση. Είπα το Θηνό που θα μια νέα στρατηγική. Καλό θα ήταν να γίνει και μια διαβούλευση πριν κάνετε την παρουσίαση, ούτως, ώστε να μα ακούσετε, να ξέρετε τι έχουμε να πούμε και τι θα θεωρούσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σα βλέπω εδώ. Ευχαριστώ, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την κυρία Ρέντινγκ. Χαίρομαι που είναι εδώ. Έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε σήμερα απόψεις και γνώμες. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Δεν θέλουμε οι να πείσουμε τους δε για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διαφοράς της αμοιβή ανδρών και γυναικών. Σας διαβεβαιώνω, κυρία Πρόεδρε, ότι γίνονται πολλές συζητήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα αναλήψεως πρωτοβουλίας και να ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης σε χώρες όπου η μισθολογική διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Αυτό ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να παραμείνει και θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Προτίθεστε να προτείνετε νομοθεσία σχετικά με το θέμα, διότι τα διαθέσιμα εργαλεία δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Άλλο ερώτημα. Η βία η απόφαση του ΕΠΣΚΟ είναι ρεαλιστική. Θα προταθεί νέα οδηγία όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας καδών γυναικών. Είχα και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα δώσω το λόγο και στο... Μάλλον θα παραχωρήσω τη θέση μου και στους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Μπάουερ. Το λόγο έχει η κυρία Νίμπλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την ευχαριστήσω ε, αφενός που μπορούμε να έχουμε εδώ τον δομημένο διάλογο αλλά και επειδή ε, δίνεται τόση σημασία στην πολιτική ισότητα. Υποβάλατε ήδη στις 5 Μαρτίου τον χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Το βρίσκω αυτό εξαιρετικό και θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, κυρία Επίτροπε. Καταρχήν, ε, στην εισαγωγή σας αναφέρατε τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να αναφερθώ στο θέμα αν στην οικονομική ζωή ε, Σκοπεύεται να εισάγετε ποσοστώσεις. Ε, στην Νορβηγία υπάρχει ποσόστοση γυναικών εδώ και αρκετά χρόνια. Στο, στις κάτω χώρες ε, αποφασίστηκε στο Κοινοβούλιο. Στη Γαλλία ε, γίνεται σχετική συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχουν λάβει σχετική απόφαση οι Γάλλοι. και στην Γερμανία βλέπουμε τις έρευνες από τις αρχές της χρονιάς Στι 15 μεγαλύτερε στις 15 μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, της χώρας μας, ε, στις... στα... στα διοικητικά συμβούλια υπάρχει μία γυναίκα και ε, βλέπουμε σε συμμετοχή 2,5% σε μια εποχή που οι γυναίκες είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέσο για τις γυναίκες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι θα κάνετε εσείς πολύ συγκεκριμένα, θα υπάρξουν ακροάσεις, εξετάζετε την κατάσταση στα κράτη-μέλη, ε, τι προτάσεις υποβάλλετε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό που αναφέρεται και στο χάρτη ε, των δικαιωμάτων. Ε, βλέπουμε τις διακρίσεις ε, στην αγορά εργασίας, τη διαφορά στις αμοιβέ. θα πρέπει να υπάρξει μία λύση, ένα μέσο για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, ώστε οι γυναίκες ώστε να μην προσφεύγουν οι γυναίκε απαραίτητα σε θέσεις απασχόλησης κακοπληρωμένες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι ε, προβλέπετε εδώ. Η ανάλυση είναι σαφής, αλλά χρειάζομαι την ε, γνώμη σας πώς μπορεί κανείς να ενεργήσει πολιτικά και νομικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω μεγάλη ικανοποίηση από τα όσα μας είπε η κυρία Ρέντινγκ. Κυρία Ρέντινγκ, όταν διεξήχθη η ακρόαση των επιτρόπων, σε αυτή την επιτροπή ανήσυχη. Δεν θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει επίτροπο όπου θα είναι τόσο αφοσιωμένη σε θέματα γυναικών. Και τώρα βλέπω ότι εσεί είστε εκείνοι που περιμέναμε για να προωθήσει το θέμα και τα πηγαίνετε πολύ καλά. Ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ μαζί μας. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία είναι λίγο αρνητική, θα ξεκινήσω από αυτή. Όσον αφορά τη βία βάση των φίλων, το συζητήσαμε αυτό, κάναμε πρόταση οδηγία, είχαμε ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί νομικά μέσα. Και δεν βλέπω τίποτα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Αναφέρεται στη χάρτα, όπως είπατε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περαιτέρω τα νομικά μέσα που ίσω να διαθέσει η χάρτα για περαιτέρω δράση που θα μπορούσε να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, μιλ... μιλούσαμε για τη ισότητα των φύλων και τη διαφορά αμοιβή των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα μπορούσαν να αναλυθούν κάποιε θετικέ δράσει, διαδικασίε, ε, εκστατείε ευαισθητοποίηση για να προωθούνται οι γυναίκε σε ηγετικές θέσεις, επιχειρήσει επιχειρήσεις και στον πολιτικό κόσμο. Θα πρέπει να πιεστούν οι χώρε να ευθυγραμμιστούν αλλά ίσως η πίεση αυτή δεν αρκεί. Αν οι μεγάλες εταιρείε θέλουν να έχουν ε, γυναίκες ε, σε υψηλές ε, θέσεις, πού θα τις βρουν. Πρέπει να κάνουμε εκτρατή ενημέρωσης. Και τι ιδέες έχετε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ για την παρουσία σας εδώ. Φαίνεται να είστε έτοιμοι για δράση. Χαίρομαι που το βλέπω αυτό. Έχει αναφερθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Ειλικρινά δεν με νοιάζει πολύ ο χάρτης. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το πρόγραμμα εργασίας. Η δράση που αναλαμβάνετε διότι σε τέσσερα χρόνια δεν θα μας θυμούνται για ωραία λόγια σε ένα κομμάτι χαρτί. Θα μας θυμούνται για το τι έχουμε πετύχει, θα έχουμε επαρκή ε, μητρική άδεια, οι άντρες θα έχουν γονική άδεια, θα υπάρχει επαρκής νομοθεσία ε, που θα μπορεί να ε, επιτρέπει τις προσφυγές σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο. Το θέμα της γονικής άδειας είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν θα δεν θα ήμουν εδώ ε, σε μια από τις καλύτερες ε, θέσεις εργασίας ε, του κόσμου εάν δεν ήταν ο άντρας μου σπίτι να φροντίζει τα παιδιά. Και θα ήθελα πολύ να ξέρω εάν θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να το πετύχετε αυτό. Εγώ θα ήθελα τα σχετικά μέτρα να συμπεριλαμβάνονται σε μία οδηγία, αλλά μπορώ να φανταστώ τα προβλήματα που θα υπάρξουν στο Συμβούλιο Μπορεί δηλαδή να είναι απαραίτητο να υπάρχει χωριστή οδηγία. Εσείς μπορείτε να προτείνετε μια τέτοια οδηγία, θα κάνετε ό,τι μπορείτε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή για να το πετύχετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιμένες. <coughs> Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ότι όταν ήμασταν μαζί σας στη Νέα Υόρκη, η ευαισθησία σας έναντι των προβλημάτων που αφορούν τη βία μεταξύ των φίλων ήταν κάτι που με συγκίνησε. Σαν εισηγείται για την προστασία των γυναικών θυμάτων βίας μεταξύ των φίλων, ανησυχώ πολύ λόγω της παρούσης καταστάσεως είδαμε τι συνέβη στη σχετινή συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων. Όλοι έχουμε κοινούς στόχους, πιστεύω. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις γυναίκες και να καταπολεμηθούμε τη βία εναντίον τους. Υπάρχουν διαφορές στον αυτή τη στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και τα διαβήματα που θέλουμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες. Ερώτημα, ποια είναι η δική σας θέση. Μπορείτε να το εξηγήσετε λεπτομερώς. Διότι πρόσφατα ξεκίνησε η συζήτηση και προβληματισμός και υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση σας, ποιες είναι οι απόψεις σας λεπτομερώς. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι προβλέπετε για όλα τα θύματα, όχι μόνο τα θύματα βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ κυρία Πλούμ. Yeah, okay. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας, κυρία Ρέντινγκ. Δύο ρωτήσεις έχω. Η μία αφορά τη χάρτα των γυναικών και η άλλη την οδηγία και τους αυταποσχολούμενους. Όσον αφορά τη χάρτα γυναικών, όπως είπε και η συνάδελφος Ζήτα Γκουρμάιερ, αυτή ήταν μια ιδέα των γυναικών του Σοσιαλιστικού Κόμματος που ξεκίνησε πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ήταν έγγραφο εργασίας που συζητήθηκε εις βάθος με τα μέλη, με τους συναδέλφους μας. Όταν ο πρόεδρος Μπαρόσο παρουσίασε τη χάρτα των γυναικών στα πλαίσια δηλώσεώς του, εξεπλάγει με τα μάλα. Διερωτήθημεν γιατί δεν έγιναν διαβουλεύσεις με εμά, με την κοινωνία των πολιτών. Λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτή η χάρτα δεν πρέπει να αντικαταστήσει το σύμφωνο για την ε, ισότητα των φύλων, ούτε τον οδικό χάρτη, ούτε τις διεθνείς συμβάσεις, έχω ερώτηση. Τι σχεδιάζετε να κάνετε διαβουλεύσεις μαζί μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα, κράτη, με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στους ε, πολίτες μας. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα για την οδηγία περί αποσχολούμενων. Κυρία Επίτροπε, να σας ρωτήσω, εφόσον είστε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θεωρείτε ότι αν θα παραμείνουν κουσίας βάσεως τα συστήματα κοινωνικής ασφαλίσεως των συζύγων ή των συντρόφων των αυταπασχολούμενων θα καλύπτονται. Ποια είναι η άποψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πέντε συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Και επειδή θα πρέπει να έχουμε και χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις στα ενδιαφέροντα ερωτήματα που ακούσαμε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρσία τώρα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας ε, παρουσιάσετε το πρόγραμμα εργασιών σας για την ισότητα των φύλων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όλες αυτές τις ιδέες. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να αποσαφηνίσουμε καλύτερα ορισμένες από τις ιδέες αυτές. Εμείς εδώ γνωρίζουμε ότι μιλούμε για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς για το μέλλον των ε, Ευρωπαίων πολιτών, γυναικών και ανδρών. ως προς τη δημιουργία νέων οικονομικών και κοινωνικών ε, φορέων. Μήπως θα έπρεπε να τις ενισχύσουμε για να ενισχύσουμε και το 52% των κοινωνιών ε, που είναι γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε σαφέστατα και πρέπει να είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε οι πολιτικές ισότητας των φύλων ε, να είναι τμήμα ολόκληρης της πολιτικής που αφορά την πολιτική για την δημογραφική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι, δεν είναι μόνο ζήτημα συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει να μιλούμε επίσης για την ε, ανάγκη επιβολής των μέτρων μείωσης των μισθολογικών διαφορών, να αυξήσουμε το μερίδιο των γυναικών ε, στην ε, ε, οικονομική δραστηριότητα και πρέπει, για παράδειγμα, να εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οι στόχοι αυτοί να είναι ποσοτικοποιημένοι, να έχουμε και στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορούμε να ε, επαληθεύσουμε την ε, καλή εφαρμογή των μέτρων που θα λάβουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα στο πλαίσιο της, Ευρω... της στρατηγικής για το 2020. Σε επειδή και άλλες συνάδελφοι μίλησαν πριν από μένα και είπαν ήδη αρκετά, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Σε σχέση όμως με τις πέντε δράσεις που αναφέρατε κι εσείς ε, και που είναι αντικείμενο αποφάσεως του ε, ε, Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πρόταση οδηγίας για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Γυναίκες και άνδρες Ευρωπαίοι κατά της βίας. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω επίσης. Και τώρα αλλά και στο μέλλον πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία αστικού και ποινικού χαρακτήρα. Δεν γίνεται να το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει και τα ευρωπαϊκά όργανα να συνεργάζονται μεταξύ τους και πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να περάσουμε στην εφαρμογή των μέτρων των συντομότερων δυνατών. Ευχαριστώ κυρία Φικεραίδο. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Οι συνάδελφοι έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων που και εμένα με απασχολούν πολύ. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την αναφορά σας στην έκθεσή μου. Πιστεύω ότι στο θεσμικό αυτό πλαίσιο υπάρχουν δύο σημαντικές ιδέες. Την μία ήδη την αναφέρατε, τις ε, συναντήσεις που θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, ώστε κάθε χρόνο να μπορεί η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να προσπαθούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν την ε, διαδικασία ε, που θα οδηγήσει στη ισότητα, διότι δεν φτάνει να υιοθετούμε έγγραφα, θα πρέπει να βλέπουμε και πώς εφαρμόζονται στην πράξη. Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα και σημαντική πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό το θέμα της συμμετοχής των γυναικών, των οργανώσεων γυναικών, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Είτε μιλάμε για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε μιλάμε για άλλα έγγραφα. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι γυναίκες και είναι σημαντικό στις αιτήσεις αυτές συναντήσεις να συμμετέχουν. Και φυσικά θα ήθελα να ξέρω τι προτάσεις θα υποβληθούν στην πράξη σχετικά με τα θέματα αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και ε, οι ιδέες αυτές ε, να συμπεριληφθούν σε προτάσεις του Κοινοβουλίου. Δεύτερη ερώτηση. Η ανισότητα στην εργασία. Είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε τη δουλειά των γυναικών, να αξιολογήσουμε και τις δουλειές τους και μάλιστα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Υπάρχει πολλή δουλειά την οποία θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Και όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές, αλλά και όσον αφορά την πληροφόρηση και τη διαμόρφωση απόψεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πολλοί συνάδελφοι μιλάμε, μιλάνε τόσο πολύ για πολλά θέματα. Να μην τα λέμε πιο απλά. Εγώ που είμαι πιο νέα βουλευτή, θα πρέπει να δώσω το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μα σήμερα. Σα ζητώ δύο πράγματα να μα πείτε πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε για την όλη θεματική ε, που είναι επίκαιρη τώρα όσον αφορά τι ηλικιωμένε γυναίκε που είναι μόνε του, κυρίω υπό το φω τη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση και μετά. Προσωπικά είμαι αντίθετη με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Γυναικών, γιατί πιστεύω ότι είναι μια επανάληψη τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή ε, Ενώσεω που ήδη ισχύει. Και αν πολεμάμε εμείς για την ισότητα των φίλων και για το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου όντω, αυτή η κάρτα, χάρτα κατά την άποψή μου είναι απλώς κάτι που δείχνει την αδυναμία των γυναικών, υπογραμμίζει την αδυναμία των γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Τρεις ερωτήσεις πάρα πολύ γρήγορες. Ε, πρώτα απ' όλα Όσον αφορά τη στρατηγική, ευχαριστώ την Επίτροπο Ρέντινγκ και πιστεύω ότι έδωσε τουλάχιστον κάποιες ενδείξεις, όμως θα πρέπει να συζητηθούν με την Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο αυτές οι προτάσεις. Όσον αφορά την Ευρώπη 2020, έχω δύο ερωτήσεις. Οι νέες γυναίκες δεν αναφέρονται πολύ συχνά. Το θέμα της ανεργίας και τη ανασφάλισης εργασία αφορά κυρίως τις νέες γυναίκες. Χρειαζόμαστε αυτό το έγγραφο αυτό να το υπογραμμίζουμε πολύ περισσότερο και αν θεωρείτε νέες μορφές ίσω ίσως και ελάχιστε ποσοστώσει εισαγωγής αυτών των ατόμων ε, στο όλο θέμα της απασχόλησης και της πράσινης οικονομίας και των δεξιοτήτων που πετούνται και σε όλες τις νέες μορφές δυνατοτήτων εργασίας δεν πρέπει να προβλεφτεί. Ένα νέο welfare κοινωνικός τρόπος απόσβεσης των συνεπειών των κοινωνικών. Να μπορούν να έχουν παιδιά οι γυναίκες, όχι απλώς να μπορούν να συμφιλιώσουν οικογενειακή και εργασία και οικογενειακή ζωή. Και να υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αφορά το ελάχιστο εισόδημα. Αυτό το ανέφερε και η κυρία Φιγκερέιδο και πολλοί από εμά στην Επιτροπή Εργασία. Μετά η συνεργασία για την ανάπτυξη. Άκουσα πολύ λίγο να αναφέρεται η αλληλεγγύη με τι χώρε, με τι γυναίκε τρίτων χωρών θα υπάρξει η δράση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν πάει, αντιπροσω... πριν πάει η αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, ε, εγώ είχα πει αν η Ευρώπη θα μπορεί να υποστηρίξει ένα αίτημα από πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις διεθνείς. Να ζητηθεί για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις των Αφρικανών γυναικών να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και την ε, προστασία των γυναικών γιατί να μην στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Ευχαριστώ για όλα αυτά. Πολλές ερωτήσεις ε, υπευλήθησαν και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ, ε, ούτως ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ. πολλοί από τους ομιλητές ε, έθεσαν τα ίδια ζητήματα, οπότε νομίζω ότι θα μπορέσω να απαντήσω αρκετά σύντομα. Θα ήθελα να αρχίσω από τη χάρτα των δικαιωμάτων των γυναικών, γιατί πολλές φορές αναφέρθηκε. Και κάποιο το είπε και σωστά, ναι, είναι μια δήλωση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, που γίνεται με οριζόντιο τρόπο μια δήλωση υπέρ των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, από τη δήλωση αυτή θα προκύψει σχέδιο δράση, στρατηγική, όπως και να το αποκαλέσει κανείς. Θα προκύψει κάτι, αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Και θα το έχετε στη διάθεσή σας στο φθινόπωρο. Θα αρχίσει λοιπόν μια πραγματική συζήτηση, θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, θα αρχίσουν ε, ε, οι έπαινοι, θα αρχίσουν οι κριτικές. Εν πάση περιπτώσει είναι μια στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει βασικά στοιχεία για το πώς θα συνεχίσουν οι πολιτικές μας. Όσον αφορά τις διαφορές στην αμοιβή, τι κάνουμε επ' αυτού. Στη στρατηγική το θέμα αυτό και η δράση που θα πρέπει να αναλάβουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό θα συμπεριληφθούν. Πρέπει να αποφασίσουμε Θέλουμε έναν υπιότερο τρόπο. Θέλουμε να νομοθετήσουμε. Να δούμε και τι δυνατότητες έχουμε, νομοθεσίες έχουμε. Μία νομική βάση για τις ποσοστώσεις, για παράδειγμα. To ask um, ourselves. Όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, θα πρέπει να τις εξετάσουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε. Το reporting στις εταιρείες, ε, διαφάνεια των αμοιβών, ε, ουδετερότητα των φύλων, όλα αυτά τα ε, μέτρα που, αναλαμβάνουμε που λαμβάνουμε ως προς την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σωστά, αποτρέπουν κακές πρακτικές. Υπάρχουν λοιπόν πολλά, πολλές δράσεις που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε και που θα σας προταθούν βεβαίως στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής και στη συνέχεια θα πρέπει να συναντηθούμε και πάλι για να αποφασίσουμε ποια, ποιες ε, στρατηγικές θα ακολουθήσουμε και ποιο θα είναι το πρόγραμμα δράσης μας, το πρόγραμμα ε, εργασίας μας για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς. The question of... Το ερώτημα τώρα, της, ε, το ζήτημα της βίας. Ξέρετε, ήδη από την ακρόασή μου πάρα πολύ σαφή όσον αφορά το θέμα της βίας και είχα πει ότι θα είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ότι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό με έναν τρόπο περιεκτικό. Θα υπάρξει ένα περιεκτικό πρόγραμμα καταπολέμησης της βίας το γεγονός ότι είμαι επίτροπος δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι επανέρχομαι σε αυτό που, είπε, σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ε, η χάρτα για τα δικαιώματα των γυναικών ε, μπορεί να συμπεριλάβει τα πάντα, το, τα θέματα της Στοκχόλμης για παράδειγμα. Πάρα πολλά ζητήματα, τι μπορεί να γίνει για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και πολλοί επίτροποι θα το λάβουν και εκείνη υπόψη. Δεν θα γίνουν λοιπόν μόνο σε μία ε, επιτροπή τα πάντα. Αυτό προσπαθούμε να πούμε στη χάρτα ότι όπου μπορούμε να αναλάβουμε δράση προς αυτή την κατεύθυνση θα το κάνουμε. Σας έδωσα ας πούμε το παράδειγμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Εγώ προτείνω να, να το εναρμονίσουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας έναν ορισμό του τι θα πει ε, αγροτηριασμός των γεννητικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης Όλες αυτές τις πολιτικές λοιπόν ε, πρέπει να τις ε, συγκεντρώσουμε κάπου. Θα υπάρχει στη στρατηγική οδικό χάρτη, όπως θέλετε πείτε το, θα, τους, ε, θα, τις, θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα μέτρα και άλλοι επίτροποι μπορεί να θέσουν να υποβάλουν ορισμένες προτάσεις. Αυτό είναι το καινούριο. Όσον αφορά τώρα την στρατηγική για το 2020, αναφέρονται πολύ σοβαρά τα ζητήματα της ισότητας των φύλων. Και η στρατηγική, ο δικός χάρτης, θα είναι ουσιαστικά η παγίωση, η εδραίωση αυτής της αναφοράς. Πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Γιατί τώρα μόνο μία ε, επισκόπηση έχουμε του, της στρατηγικής του 2020. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής υπάρχει ας πούμε, με αυτό ασχολείται και η Επιτροπή των ε, Κοινωνικών ε, Θεμάτων και Απασχόλησης, που είναι επίσης συναρμόδιοι για αυτό που κάνουμε. Υπάρχει και ένα ζήτημα αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο Επίτροπος ή ε, η Επίτροπος για την αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει επίσης να ε, μας βοηθήσει. Αν τα λάβετε όλα αυτά υπόψη, θα καταλάβετε ότι είναι μια δήλωση πίστεως ε, η χάρτα των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, δεν αφορά μόνο το χαρτοφυλάκιο των δικαιωμάτων των γυναικών. Όχι. Και οι υπόλοιποι επίτροποι πρέπει να υποβάλουν τα δικά τους, τη δική τους άποψη για τα, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα στα σημαντικότερα ζητήματα. Το μόνο που μένει είναι η εντολή προστασίας. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα. Όλοι πιστεύουν και όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των γυναικών από τη βία. Το θέμα είναι ότι τα μέτρα έχουν τόσο άσχημα προετοιμαστεί που η πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι κατά. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είχε αντιρρήσεις. Πάρα πολύ ε, νομικοί είπαν ότι ε, είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί βεβαίως θα έχουν δουλειά έτσι. Πρόκειται για κάτι που ε, ουσιαστικά θυματοποιεί τα θύματα δεύτερη φορά. Γι' αυτό έλεγα να μην το προωθήσουμε αυτό το θέμα. Στο τελευταίο Συμβούλιο ε, Υπουργών Δικαιοσύνης οι περισσότεροι υπουργοί είπαν να μην συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, δηλαδή να ξαναρχίσουμε από την αρχή για να έχουμε ένα ε, καινούριο κείμενο το οποίο δεν θα δημιουργεί, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα αλλά θα επιλύει αυτά που υπάρχουν. Κάτι πιο συγκεκριμένο εν πάση περιπτώσει. Να είναι μια πρωτοβουλία για παράδειγμα στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Κάτι που δεν θα μας πάει... Δεν μπορούμε να, να, να το κάνουμε αυτό ε, εις βάρος των γυναικών. Εγώ αυτό που είπα είναι να ξεχάσουμε αυτό που έχει γίνει ως τώρα, να ξαναρχίσουμε τη διαδικασία από την αρχή. Στις 25 Μαΐου θα συναντηθούν οι εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό, προκειμένου να δούμε, να βρούμε μία λύση. Η λύση ενδεχομένως να είναι νομοθεσία που να αφορά αρχικά μόνο τις γυναίκες, μια μικρότερη εμβέλεια νομοθεσία και μετά στι αρχέ του 2011 να έχουμε ένα ευρύτερο πακέτο που θα συμπεριλάβει ε, και διοικητικά ζητήματα, ιδιωτικά ζητήματα. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν ποινικοποιήσει όλα τη βία κατά των γυναικών. Μπορεί να σας αρέσει αυτό ή να μην σας αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι διοικητικό μέτρο σε κάποιες χώρες, όπως στη δική μου χώρα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τα ποινικά μέτρα να τα μπερδεύουμε με διοικητικά μέτρα. Και αυτό σας το λέω για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και να το κάνουμε καλά, με τέτοιο τρόπο που να βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων των και συμφωνώ με όλους όσους είπαν ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες, εντάξει το 90% μπορεί να είναι γυναίκες, ε, να είναι, να είναι γυναίκες τα θύματα, αλλά συχνά είναι και παιδιά και άντρες. Όλο και περισσότερο το βλέπουμε αυτό. Οπότε, Α το επεξεργαστούμε όλοι μαζί. Κρίμα που έγιναν έτσι τα πράγματα. Εγώ πραγματικά πολύ λυπάμαι. Πρέπει να είχαμε κάνει μια σοβαρή μελέτη αντικτύπου. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αν υπουργοί ε, συγκεντρωθούν, συμφωνήσουν και κάνουν μια πρόταση, δεν χρειαζόμαστε μελέτη αντικτύπου και βλέπετε το αποτέλεσμα. This is very serious. Δεν είναι αστείο λοιπόν. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα και πρέπει να έχουμε και μια σοβαρή βάση για να το ε, επιλύσουμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση να τοποθετηθώ. Και όπως σας είπα, η πρότασή μου θα γίνει στις αρχές του 2011 με ένα ευρύτερο περιεκτικό πακέτο αντιμετώπισης των προβλημάτων των θυμάτων, όχι μόνο της σεξουαλικής βίας, αλλά και θυμάτων άλλων. Κάποια μέτρα είναι ποινικά, κάποια μέτρα μπορεί να, ε, ε, να χρειαστεί να βοηθήσουν ε, και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, η ανάλυση έχει δρομολογηθεί και οι σχετικές δράσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε υγιή νομοθεσία που δεν θα μας πάει στο δικαστήριο. Εκ μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο Ρέντινγκ για τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινέ μας εργασίες για θέματα ισότητας. Να ευχαριστήσω θερμά την ε, κυρία Ρέντινγκ που συμμετείχε στη συνεδρίασή μας σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, να συνεχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ. Please. Παρακαλώ, πρέπει να ξεκινήσουμε διότι έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια του πρωινού. Προχωράμε δηλαδή στο θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η εντολή για, για τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Η κυρία Καρσία Πέρες, η συγκήτρια, έχει έτοιμα γνωμοδότηση και καθότι η Κομισιόν μόλις στις 27 Απριλίου υπέβαλε την πρότασή της, και καθότι η Επιτροπή μας έχει τη δυνατότητα να συντάξει γνωμοδότηση ε, στην, ε, στην ε, αρμόδια επιτροπή πριν την ψηφοφορία της τη 2η Ιουνίου έχουμε εφαρμόσει σύντομη διαδικασία. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν η 13η Απριλίου. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό μόνο στα αγγλικά. Δεν έχουμε συζητήσει νωρίτερα το θέμα αυτό. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα για μια σύντομη συζήτηση πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Καρσία Περές. Χαίρομαι που η εισηγήτρια σε τόσο, η συντάκτρια σε τόσο, χρονικό, σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να συντάξει μια γνωμοτότηση. Παρακαλώ, κυρία Γκαρσία Πέρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Τονίζω πρώτα απ' όλα ότι όσον αφορά τη διαδικασία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει αυτό το θέμα, αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όπου το Κοινοβούλιο γίνεται πραγματική αρχή του προπολογισμού όσον αφορά τον, την κατάρτιση του προπολογισμού χάρη στη συνθήκη τη θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στι θέσει μας. Και θα πρέπει επίσης να είμαστε σοβαροί στη δουλειά που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν σοβαροί κατά το παρελθόν. Αλλά κατά το παρελθόν δεν είχαμε αρκετό χρόνο ούτω ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν οι συνάδελφοι τα διάφορα σχόλιά τους εκτενώς. Θα συνεχίσουμε να σχολιάζουμε όποτε έχουμε την ευκαιρία, όπως να υπάρχουν αναγκαίοι πόροι για τα διάφορα προγράμματα που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών, για το πρόγραμμα Δάφνη για τη χρήση των διαθωτικών ταμείων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της ισότητας των φύλων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μπορεί να δρομολογεί διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες πρωτοβουλίες να βοηθούν τις γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να διατίθενται και επαρκή πόροι για πρωτοβουλίες του τύπου e-progress, ούτως ώστε να μην μειώνονται οι πόροι και επίσης και διάφορα συναφή θέματα αυτά που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Καταφέραμε λοιπόν εδώ να δώσουμε μια γενική εικόνα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες, τους ευχαριστώ που κινήθηκαν γρήγορα. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε λεπτομέρειες τροπολογίες αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν παρατηρήσει για το θέμα αυτό. Εάν όχι, να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόλαντ από την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το ψήφισμα, έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλετε να απευθύνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλετε να σας παρουσιάσουμε το σχέδιο προπολογισμού. Det vore intressant för utskottet om vi kunde... Θα ήταν ενδιαφέρον για την Επιτροπή αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με την ε, πρόταση αυτή για τον προϋπολογισμό που αφορά την Επιτροπή μας. Αν είναι δυνατόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόλαντ και πάλι, παρακαλώ. Oui, euh, <coughs> ναι, λοιπόν, είμαι στη Γενική Διεύθυνση την υπεύθυνη για την απασχόληση μπορώ να μιλήσω για αυτές τις πτυχές που ανέφερε και η συγγήτρια. Για το πρόγραμμα Progress, όταν υιοθετήθηκε το πρόγραμμα μικροχρηματοδότηση έγινε μια δήλωση. Έλεγε ότι αν υπάρχει επαρκές δημοσιονομικό περιθώριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς να το πω, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τα επιστρέψει τα 5 εκατομμύρια στο Progress. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το σημείο για την ισότητα των φύλων στα διαθετικά ταμεία. Είναι κάτι που προγραμματίστηκε, ελέγχεται, παρακολουθείται προσεκτικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τα κάτι μελη Διάφορες αξιολογήσεις διεξήχθησαν προς αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο η διάσταση ισότητα των φύλων λαμβάνεται υπόψη θετικά ταμεία και πιο συγκεκριμένα στο κοινωνικό ταμείο όσον αφορά το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων θα είναι αυτόνομο από τον μήνα Ιούνιο και, και μεταξύ του Ινστιτούτου αυτού και των ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατεβλήθησαν προσπάθειες για να ξεκινήσουν δραστηριότητε ε, εγκαίρως. Όσον αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, δεν εξαρτάται από Γενική Διεύθυνση για την απασχόληση, οπότε δεν μπορώ να σα δώσω σχετικέ πληροφορίε. Αυτά. Λυπάμαι. Ε, μπορώ να απαντήσω σε πιο συγκεκριμένε ερωτήσει, αν αυτό επιθυμείτε. Σα ευχαριστώ πολύ για τι πληροφορίε αυτέ. Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε τι ψηφοφορίε. Θα ξεκινήσουμε με τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. 15 voting. 15 υπέρ, 14 κατά. Να ξαναψηφίσουμε, διότι αρκετοί δεν ψήφισαν. Αρχή της ψηφοφορίας, παρακαλώ ψηφίστε. The vote Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγ... ε, απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ε, χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Αρχή της ψηφοφορίας. Πρώτο μέρος. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 13 κατά. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 6. Λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται 16 υπέρ. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ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 Η 14 απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. πού. Thanks, Mrs. Luling. Κυρία Λούλινγκ, ευχαριστώ. Ωραία, προχωράμε στην επόμενη ψηφοφορία ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Έχουμε συζητήσει την, ε, την έκθεση αυτή επανειλημμένα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λούλινγκ που έχει εργαστεί με μεγάλη αφοσίωση πάνω στο θέμα αυτό. Μετά την έγκριση στην Επιτροπή μας, έχουμε εντολή διαπραγμάτευσης ε, για μια ομάδα ε, της οποίας ηγείται η κυρία Λούλινγκ, η συγγήτριά μας. Ε, η ομάδα αυτή θα διαπραγματευτεί με, την, με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να προσπαθήσει να καταλήξει σε λύση κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Δίνω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ. αν έχει παρατηρήσεις πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ κυρία Λούλινγκ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω όλου του εισηγητέ και οι όδη εισηγητέ, επίση και τα μέλη, για την συνεισφορά του, για τι προσπάθειε που κατέβαλαν του, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να τεθεί σε ισχύ επί Ισπανικής Προεδρίας. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία, κυρίως τον κύριο Κάρλος Γκαρσία, Κορταζάρ και τον του, τους συναδέλφους του που έκαναν τιτάνιο έργο ε, για να προσπαθήσουν να πείσουν το Συμβούλιο να ενστερνιστεί σε πρώτη ανάγνωση σειρά τροπολογιών μας και τις τροπολογίες μας για τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση. Εγώ πιστεύω ότι άνευ της εργασίας τους, της αφοσίωσής τους, δεν θα το πετυχαίναμε αυτό και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοήθησε πάρα πολύ, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο, το οποίο κείμενο θα μπορεί να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα ήθελα, κυρία Προέδρε, να ζητήσω να δώσετε εν συντομία το λόγο στον κύριο Κορταζάρ της Ισπανικής Προεδρίας για να σας εξηγήσει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Λούλινγκ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοτζάρ από την Ισπανική Προεδρία. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Ιστορική δυνατότητα θα έλεγα που μου δίνετε μετά από κάποιες συναντήσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, επί τη ευκαιρία της τελευταίας οδηγίας για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, ετέθη το θέμα της το και κυρίως υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις από Συμβουλίου, υπήρχαν δισταγμοί όσον αφορά την έγκριση νέων μέσων και εργαλείων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει αυτό το μέσο που συζητούμε. Πιστεύω ότι χάρη σε αυτό το μέσο ανοίγουμε ένα μονοπάτι πάρα πολύ σημαντικό προς συμφωνίες, προς μια Ευρώπη κοινωνική, προς μια Ευρώπη ισότητας. Ίσως το κείμενο του Συμβουλίου που θα τροποποιηθεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην είναι το καλύτερο κείμενο στον κόσμο, αλλά είναι το καλύτερο εφικτό κείμενο. Αυτό σας το λέω σταθμίζοντας τα λόγια μου. Δεν είναι το καλύτερο κείμενο του κόσμου, δεν είναι το κείμενο που το Συμβούλιο θα επιθυμούσε να έχει, αλλά είναι το καλύτερο δυνατόν, διότι μας επιτρέπει να κάνουμε γιγάντιο βήμα όσον αφορά την προστασία των αυτοαπασχολούμε των εξαρτήτων εργαζομένων. Προβλέπεται ε, ε, άδεια μητρότητας 14 εβδομάδων και περνά αυτό το μέσο επίσης στην κοινωνική, μέσω της κοινωνικής ασφαλίσεως και περνάμε και στην αναγνώριση των περιστατικών που οδηγούν σε αυτή τη χορήγηση. Και από την πλευρά μας και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι επιδείξαμε ρεαλισμό διότι από ό,τι κατάλαβα η Επιτροπή σας υποχώρησε εναντί ε, του ρεαλισμού που θεώρησε ότι είναι σημαντικό να επιδειχθεί. Είναι μια οδηγία που μπορεί να αποτελέσει τη ρίζα μελλοντικών οδηγιών. Είναι γιγάντιο το βήμα που κάνουμε σήμερα. Και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της οδηγίας που ελπίζω θα μπορέσει να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αν όλα πάνε καλά, στην Κορεπέρ της Τετάρτης 12 της Μαΐου. Εάν ε, υιοθετήσετε κάποιες τροπολογίες εδώ, το κείμενο θα μπορέσει να εγκριθεί και να σας υποβληθεί και πάντα υποθέτοντας ότι θα μπορέσετε να το υιοθετήσετε στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 18 του μηνός. Ευχαριστώ την κυρία Λούλινγκ για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Εν πάση περιπτώσει από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι η Ισπανία έμαθε πολλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η κυρία Λούλινγκ ήταν δασκάλα σε αυτό το τομέα, μας καθοδήγησε ε, για να καταλήξουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα έχουμε ένα κείμενο συνενετικό στις 18 Μαΐου που θα συμφωνούν όλα τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι είμαι σκιώδης εισηγήτρια και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούλιν για την συνεργασία, να ευχαριστήσω και την Ισπανική Προεδρία, τον κύριο Κάρλος Καρσία και τον βοηθό του. Μπορεί πράγματι να μην πρόκειται για το καλύτερο δυνατό κείμενο. Θέλαμε όμως να προχωρήσουμε και να υιοθετηθεί αμέσως το κείμενο, διότι χρειαζόμαστε κοινωνική προστασία και νομοθετική ρύθμιση για όσους ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και τους ε, εταίρους τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της παρούσας οικονομικής ε, κρίσης ακόμα και αν η οδηγία αυτή εφαρμοστεί σε τρία χρόνια από τώρα. Όσον αφορά την τροπολογία 28 στον κατάλογο των ψηφοφοριών, θα ανακοινώσω την πρόθεσή μου. Αυτή είναι η διαδικασία ή μου επιτρέπετε να το πω τώρα. Ε, να το κάνω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κατάλαβα ότι η τροπολογία μου, η παριθμόν 28, έχει να κάνει με την υιοθέτηση της, ε, της οδηγίας αυτής στο Συμβούλιο. Αποφάσισα λοιπόν να αποσύρω την τροπολογία 28, αλλά επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να την επανυποβάλλω στην Ολομέλεια, εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με το Συμβούλιο μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αυτή είναι η απόφασή μου. Διότι δεν θέλω εγώ να προκαλέσω μπλοκάρισμα της οδηγίας αυτής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ανακοίνωση της κυρίας Πλούμ σχετικά με την τροπολογία 28. Δεν θα ξεκινήσουμε πάλι τη συζήτηση, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 αποσύρθηκε από ό,τι ακούσαμε. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 αποσύρεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 αποσύρθηκε. Η 32 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε την 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 αποσύρθηκε. Η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε την 14. Έχουμε προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει ε, ω στην την προφορική τροπολογία. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ της 14 κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 1 και τη 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 16 αποσύρθηκε. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 4 και την 17. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 19 και 5 αποσύρονται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 καταπίπτει διότι υιοθετήσαμε την 18 και το ίδιο ισχύει για την 20. Ε, 22 αποσύρεται. 6 δεν πρέπει να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε τώρα την 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Λυπάμαι κυρία Λούλινγκ. Απορρίφθηκε η τροπολογία. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 αποσύρεται και 28 δεν ψηφίζεται. Οι 8 και 26 δεν ψηφίζονται. Έχουμε λοιπόν την, οριστική, την τελική ε, ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά. Λήξη της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι 29 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Λούλινγκ. Την ευχαριστώ για τη δουλειά της. Προχωράμε γρήγορα στην επόμενη ψηφοφορία. Το θέμα είναι η αξιολόγηση του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Φιγκερέιδο, για σύντομη παρατήρηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο μου σχόλιο είναι να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν ε, στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Η συμβολή σας ήταν πολύ σημαντική. Πολλά, πολλοί ευρωβουλευτές ε, υπέβαλαν προτάσεις ε, και οι σκιώδεις εισηγητές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πολιτικές ομάδες ε, συνεργαστήκαμε όλοι πολύ καλά για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες έχουμε για τη συγκεκριμένη έκθεση και αυτό είναι το, αντικείμενο, αυτό είναι το αποτέλεσμα σκληρή δουλειά που κάναμε όλες τι προηγούμενες συνεδριάσεις. Επίσης είχαμε και ε, κάποιες ε, κατηδίαν ε, επαφές και το αποτέλεσμα ήταν οι τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες που σας είπα. συμβιβασμού μεταξύ των ευρωβουλευτών ε, από διάφορες πολιτικές ομάδες και θα θέλα και πάλι να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Δεν συμφωνούσαμε πάντα για όλες τις πτυχές της έκθεσης αυτής και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ε, διαστάσεις απόψεων, θα το δείτε και στον κατάλογο της ψηφοφορίας, αλλά κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι διακυβεύεται το, η ουσία, του, το περιεχόμενο της έκθεσης λόγω της ε, διάστασης των απόψεων. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή μας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι μία ακόμη πτυχή υπάρχει που δεν καταφέραμε να επιλύσουμε και βέβαια θα τεθεί σε ψηφοφορία τώρα το ζήτημα αυτό. Εννέα τροπολογίες υπέβαλα εγώ ίδια. Θα τις ψηφίσουμε. Και όλα αυτά με σκοπό να υπάρξει συνένεση στο πλαίσιο της Επιτροπής μας Βελτιώνω λοιπόν, τροποποιώ τη δική μου την έκθεση με σκοπό τη συνένεση. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για την έκθεσή μου. Η κυρία Ρέντινγκ ε, τόνισε ορισμένες πτυχές που είναι σημαντικές και για τη συγκεκριμένη έκθεση. Νομίζω ότι στην Ολομέλεια θα υπάρξει συνένεση για την έκθεση αυτή και νομίζω ότι το αποτέλεσμα της επερχόμενης στρατηγικής θα είναι επίσης θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φιγερέιδο. Παρατήρηση από την κυρία Γκουμάη, παρακαλώ να πω κάτι. Έγινε σκληρή δουλειά. Πολύ σημαντική έκθεση. Ήταν ευκαιρία να συναντηθούμε και να καταλήξουμε βιβασμούς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις συμβαστικές λύσεις. Έχουμε σαφείς συστάσεις για το μέλλον. Για τον επόμενο δικό χάρτη ή όπως άλλος αποκλειθεί, η οπως αλλος αποκληθεί Ρέντινγκ θα συνεργαστεί στα σοβαρά μαζί μας. Ευχαριστώ εκ νέου για τη συνεργασία. Ευχαριστώ και τον Ζόλταν ιδιαίτερος. Έκανε πάρα πολλή δουλειά προσπαθώντας να φέρει σε επαφή όλες τις γυναίκες μεταξύ τους για να συνεννοηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ρωτώ αν μπορούμε να ψηφίσουμε on block, όλες μαζί δηλαδή, τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπορούμε? Ναι, όχι. Ωραία. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου δεν ακούσαμε. 2, 3, 4, 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Ε, συγγνώμη, για την 65 έχουμε προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. 65 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 15 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε στην 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 74 καταπίπτει, 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Να ελέγξουμε την 147 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, εντάξει. Αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 90. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. 91. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 και 95 καταπίπτουν. Προχωράμε στην 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ε, ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την 96. Λήξη της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε στην 102 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας, 102 το πρώτο μέρος. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 7 κατά. Δεύτερο μέρος ε, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας ψηφίσουμε την 101. Λήξη της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας ψηφίζουμε την 109. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 κατά, 13 υπέρ. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήταν πολύ σαφές. Μπορούμε να ψηφίσουμε στην 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας 114. The vote is closed. Ε, adopted 16 in favor. 16 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 119 αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 11 κατά. 120 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 και 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 135 καταπίπτει όπως και η 136 προχωράμε στην 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε αρχή της ψηφοφορίας 137 Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε.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 13 την καταψήφισαν. Προχωράμε στην 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 18. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 13 κατά. Προχωράμε στη συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και προχωράμε στην 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 21. Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. Περνάμε στην 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27. Να ελέγξουμε την 26. Αρχή της ψηφοφορίας. Τροπολογία 26. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 κατά, 13 υπέρ. Πάμε στην 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, α, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. «37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και τώρα συνάδελφοι, έχουμε την τελική ψηφοφορία. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 2 κατά, 11 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Φιγερέιδο. Ευχαριστώ. Προχωράμε τις ψηφοφορίες. Προχωράμε στο θέμα της σημερινής διάταξης υπαριθμών 13, όπου η συγητής είναι ο κύριος Ρωμέβα. Πρόκειται για τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δίνω το λόγο στην κυρία στον κύριο Ρώμεβα. Στον κύριο Ρώμεβα πριν ε, την ψηφοφορία για μια σύντομη ε, θα είμαι πολύ σύντομο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί της ουσίας. Έχουμε πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες και καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο, στο οποίο εκπροσωπούνται λίγο πολύ όλες οι πολιτικές ομάδες. Όλες οι τροπολογίες σκοπό είχαν ένα συνενετικό κείμενο και ελπίζω ότι θα σας ε, βρουν σύμφωνους ε, οι τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, eh, ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Α, η κυρία Λούλινγκ θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ απέσυρα κάποιε από τις τροπολογίες ε, που είχαμε υποβάλει από κοινού με την κυρία Κλα, ε, Η κυρία Κλά, βεβαίως ε, επίσης τι αποσύρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κανονισμός λέει ότι εφόσον η κυρία Κλάς έχει συνυπογράψει, θα έπρεπε και εκείνη επισήμως να αποσύρει την υπογραφή της. Η κυρία Κλάς είναι εδώ δεν μπορεί να είναι εδώ, λέει η κυρία Λούλινγκ. Μου είπε εμένα να πω ότι τις αποσύρω γιατί τις υποβάλαμε από κοινού. Το είχα πει και στον κύριο Ρωμέβα. Τι λέει ο εισηγητή γι' αυτό. Μήπω έχετε πληροφορίε από αυτό. Αποσύρονται ναι ή όχι. Ναι, γνέφει ο κύριο ε, Ρωμέβα. Οπότε αποσύρονται οι τροπολογίες και της κυρίας Λούλινγκ και του, και, και της κυρίας Κλάς. Ναι, λέει ο κύριος Ρωμέβα, εμεί δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εφόσον η κυρία Λούλινγκ λέει ότι αποσύρονται οι τροπολογίες οι δικέ τη που τι είχε υποβάλει από κοινού με την κυρία Κλάς, εγώ τι μπορώ να πω. okay, då beslutar vi att ehm, de ändringsförslag Λοιπόν, άρα αποφασίζουμε ότι αυτές οι δύο τροπολογίες έχουν αποσυρθεί από την κυρία Λούλινγκ και από την κυρία Κλάς. Ωραία. Μιλάμε για την 57, 74, 78, 79... 82, 120, 123 και 137. Αυτές είναι οι τροπολογίες που έχουν αποσυρθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Α, καταπίπτει. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορία για την 53. Πέρα της ψηφοφορία. 16 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Η 54 καταπίπτει, οπότε 55 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, Έλεγχος της 55. Έλεγχος της 55 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 16 προς 12. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 57 έχει αποσυρθεί όπως είπαμε. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικό στην 60 έναρξη ψηφοφορίας. Εδώ. Πέρας. Ναι, όντως ε, απορρίπτεται. 15 κατά, 14 υπέρ. 61 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 63. Α, είναι ταυτόσημη, οπότε πάμε στην 65. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε την 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο της 73 έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Ναι, όντως απορρίπτεται. 16 κατά 13 υπέρ. 74 ε, αποσύρεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να την ελέγξουμε. 76 λοιπόν, έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. 15 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78, 79 έχουν αποσυρθεί. 80 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 81 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. ήρθε. 87 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Α. Ναι, ναι, την ψηφίζουμε. Δεν έχει αποσυρθεί. 88 και 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην 90. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 12 υπέρ, 16 κατά. Άρα απορρίπτεται. 91. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Την 91. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας.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 από την κυρία Λούλιν και την κυρία Κλάς. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα και το δεύτερο τμήμα. Στην παράγραφο 12 λέμε. Γιατί έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Άρα ψηφίζουμε τα δύο τμήματα. Ψηφίζουμε την παράγραφο 12, όχι την τροπολογία 92. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία, αλλά η παράγραφος 12 εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει να την ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Και αυτό μας το ζήτησε η ομάδα των συντηρητικών. Άρα, ψηφίζουμε την παράγραφο 12, το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 93. Όχι. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την 95 την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Έναρκη, έναρξη ψηφοφορίας για την 95. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. 16 κατά 12 υπέρ. 96. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 97. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται όντως 16 υπέρ 12 κατά. Συμβιβαστική υδροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρι... Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Γιατί 98 εγκρίθηκε ήταν στο συμβιβασμό, στη συμβιβαστική τροπολογία. Οπότε πηγαίνουμε στην 104 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει και αυτή, λέει η πρόεδρος. Καταπίπτει και 104. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εντάξει κυρία Γιανακουδάκη. 105 λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. 15 κατά 13 υπέρ. So we go to... Περνάμε στην 106. Είδα. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Της 106. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λάθος έκανα. Ε, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 108 καταπίπτει. 109. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Λοιπόν, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 117. Πέρα. 11 υπέρ 16 κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 120 έχει αποσυρθεί. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 αποσύρεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται την ελέγχουμε όμως και ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας 127 την 127 ψηφίζουμε. Yes, we come back to that. Now we have vote on 127. Ψηφίζουμε την 127, την ψηφίσαμε πέρα τις ψηφοφορίες και την απορρίψαμε. 15 κατά 13 υπέρ. 56, no. That's, uh, no. No, no, now it's 126 uh, can be put to, there was an agreement with. 128. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος της 138. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 21 κατά και 6 υπέρ, άρα απο, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος της 144, έναρξη ψηφοφορίας. The vote Πέρας. Απορρίπτεται 16 προς 12. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. Έλεγχος. Εντάξει. Έλεγχος τροπολογίας 1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 16 κατά 12 υπέρ. Άρα απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος της τροπολογίας 8. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 προς 13 λέει η πρόεδρος. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, ε, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος της 20 έναρξης ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. Δεκατρία, δεκατρία και μία αποχή. Άρα απορρίπτεται. 21. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κα, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται. Και πηγαίνουμε στην 29 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά απόχέ. απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 27 ψηφίσαντες, 25 ε, υπέρ, ε, μία, αποχή, ένα, ένα, μία ψήφος κατά και ε, μία αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια, κύριε Ρωμέβα Ιρουέβα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία τους ε, κατά διάρκεια των ψηφοφορίων αυτών που κάτσαν αρκετή όλα. Ευχαριστώ πολύ. but I want to say Thank you. Thank you, Mrs. President. Ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι αυτή η Επιτροπή είναι πολύ, πολύ σημαντική. Ασχολούμαστε με το θέμα της ισότητας των φίλων και της ισότητας των ευκαιριών. Γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ για τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής ή δυνατόν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε οι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές να έχουν διερμηνία στη μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Το ίδιο και εγώ, λέει και Σουβίρ. Εστονική διερμηνία θέλω εγώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας ε, για την διερμηνία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ε, διερμηνία και σε αυτές τις γλώσσες. Ledamöter, Συνάδελφοι βουλευτές. Please take your seat. I have Παρακαλώ καθίστε, έχω να κάνω μια ανακοίνωση σημαντική. Παρακαλώ καθίστε. Όταν αποφασίσαμε σχετικά με την ημερήσια διάταξη, προσθέσαμε ένα θέμα στο οποίο φτάσαμε τώρα. Πρόκειται για πώς θα γίνει η παρακολούθηση της συνέχειας του χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών, το follow-up δηλαδή. Πρόκειται για προφορική ερώτηση για την οποία θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ξεκινήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Ο λόγος για το θέμα αυτό, ο λόγος που θέσαμε το θέμα αυτό στην μερική διάταξη είναι ότι Όπως ακούσαμε και από την Επίτροπο Ρέντινγκ σήμερα, η Κομισιόν ε, εξόδου γνωμοδότηση για τον χάρτη των δικαιωμάτων των γυναικών ε, στα πλαίσια της ημέρας των γυναικών. Συζητήσαμε έναν χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών ε, σε, στη συνάντηση των συντονιστών μας και συμφωνήσαμε. Και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικός ένας χάρτης δικαιωμάτων των γυναικών και συζητήσαμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, να παρακολουθήσουμε την συνέχεια που θα δοθεί στη γνωμοδότηση για τον χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών. Αποφασίσαμε να προτείνουμε προφορική ερώτηση Όχι για να ζητήσουμε επίσημα να συμπεριληφθούν κάποια πράγματα στο χάρτη, αλλά για να συζητήσουμε με την Κομισιόν τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε συνέχεια στις, ε, στην πρόταση αυτή. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι πρόσφατα ψηφίσαμε σχετικά με μία τροπολογία στην, στην έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας Φιγερέιδο. Η τροπολογία έλεγε ως εξής, την επαναλαμβάνω. Επιμένουμε η Κομισιόν να συμβουλεύεται την Επιτροπή μας όταν κατά την εκπόνηση, να συμβουλευτεί την Επιτροπή μας κατά την εκπόνηση του χάρτη δικαιωμάτων των ε, γυναικών. Είναι μια τροπολογία που βρήκε την υποστήριξη της τροπολογίας κατά την ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Φιγερέιδο. Δίνω το λόγο στους βουλευτές ε, για συζήτηση της προφορικής ερώτησης. Δεν συζητάμε ψήφισμα, συζητάμε μόνο προφορική ερώτηση για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής. Η κυρία Μπάουερ ζήτησε το λόγο και κατόπιν η κυρία Γκουμάη. Πρώτα η κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω την άποψή μου επί του θέματος και ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνατε όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί στο θέμα. Μετά από τις συζητήσεις με την κυρία Επίτροπο, έχω την εντύπωση ότι έχουμε πολλές απαντήσεις για τα τεκτενόμενα. Και όσον αφορά την προφορική ερώτηση, θα έχουμε απλώς τυπικές απαντήσεις. Διότι κατέστησα φέστατον ότι δεν έχουν ακόμα τίποτα έτοιμο. Και όσον αφορά τις ερωτήσεις μας και ερωτήσεις σας, θα έχουμε ερω... απαντήσεις μόνο όσον αφορά τον οδικό χάρτη. Μετά από τις θεσινές συζητήσεις για την εφαρμογή, μετά από διήμερη συζήτηση, για το πώς θα προχωρήσουμε, in this stage it's, uh, it's, uh, it has not too much meaning to ask. Σε αυτή τη φάση δεν έχει νόημα να υποβάλουμε αυτές τις ερωτήσεις γιατί όπως σας έλεγα και λέω επανειλημμένα απλώς θα πάρουμε τυπικές απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπάουρ. και ακόμα παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω την άποψή μου. Ψηφίσαμε μια τροπολογία όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Φιγκερέιδο και ζητούμε εκεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να προετοιμαστεί μια χάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας στο μέλλον. Υπό το φως αυτών των πληροφοριών πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη θεμητή ερώτηση, την έχουμε συντάξει πολύ καλά. Αν ακούσατε την Επίτροπο, η Επίτροπος δεν παρουσίασε τον οδικό χάρτη, διότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά πιστεύω ότι ο χάρτης αυτός θα υποβληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο, πριν να μας παρουσιάσει τον οδικό χάρτη, θα έρθει μαζί μας, να, θα έρθει κοντά μας να συζητήσει. Σήμερα το πρωί πράγματι αναφερθήκαμε στη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Γυναικών με την Επίτροπο. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό να επιληφθούμε του θέματος και να δούμε τι απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν στις δικές μας ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε αυτή τη στρατηγική η διάσταση των φίλων, της ισότητας των φίλων είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν στη στρατηγική της Λισαβόνας, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα για να συνεχιστεί το mainstreaming, να συμπεριλαμβάνεται αυτή η πτυχή σε όλες τις πολιτικές. Ήταν η πρώτη επαφή με την Επίτροπο και είναι προφανές ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος μαζί της, κυρίως αφού ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλησεν. Συμφωνώ με την κυρία Μπάουερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δώσει απαντήσεις πρακτικές για το τι πρόκειται να κάνουν, αυτό θα ακολουθήσει. Το ερώτημα είναι περισσότερο διαδικαστικό, το θέμα είναι περισσότερο διαδικαστικό. Είναι η σωστή στιγμή να υποβάλουμε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πώς θα προσεγγίσουν την κατάρτιση προγράμματος ερωτήσει. Θα ήθελα να προτείνω να προσθέσουμε μία ερώτηση. ή δεν ξέρω πώς θα αποκληθεί βάσει τη χαρτα Υποστηρίζω το να τεθούν αυτές οι ερωτήσεις. Θα ήθελα να προτείνω να προσθέσουμε μία ερώτηση. Η κυρία Ρέντινγκ επανειλημμένα τόνισε ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της χάρτας είναι ότι όχι μόνο αυτοί, αλλά όλοι οι επίτροποι έχουν δεσμευθεί να τηρήσουν αυτή τη χάρτα. Άρα είναι, θα είναι πολύ σημαντικό μέσο για το mainstreaming. Διαδικαστικά όμως, πώς θα υλοποιηθεί αυτό, πώς θα το υλοποιήσουν. Ότι τα προγράμματα όλων των άλλων επιτρόπων θα αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της χάρτας, δηλαδή τους στόχους που θα περιέχει η χάρτα. Ευχαριστώ κύριε Κόνετσεν. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλης. Είναι κυρία Μωρέ, η αντιπρόεδρος κυρία Μωρέ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι υποστηρίζω τη θέση της κυρίας Μπάουερ. Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα σημαντικότατο, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε τη στατηγική για την προσέγγιση του θέματος μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρατε και μεν και δε τη στρατηγική της Λισαβόνας λέγοντας ότι η μάχη για την ισότητα των φύλων συμπεριλαμβανόταν και υπογραμμιζόταν στη στρατηγική της Λισαβόνας και τα πράγματα ήταν λιγότερο ξεκάθαρα στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Εγώ σας παραπέμπω στο εξή θέμα. Σημαίνει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ένα θέμα στην ε, στρατηγική ή ότι ζητάμε συγκεκριμένες δράσεις. Εμείς περισσότερο θέλουμε να δίνετε συνέχεια σε δύο άξονες όσον αφορά την ισότητα των μισθών και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Περισσότερο αυτό θέλουμε παρά να θέτουμε τυπικές ερωτήσεις οι οποίες θα παραμείνουν χωρίς κάποια αποτελεσματική απάντηση για την ώρα. Αυτή θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας εργασίας θα πρέπει να το αναλύσουμε το θέμα, να επιλέξουμε τους άξοντες που θα είναι φορείς αποτελεσματικότητας της δράσης. Εγώ θα πρόσεχα πάρα πολύ τους στόχους μας. Θέλουμε οι στόχοι μας να ε, ακολουθούνται από συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ κύριε Μαρία. Η κυρία Φεγκερέιδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα τα διάφορα που υπόθηκαν. Χτες συζητήσαμε επίσης το θέμα. Αυτό που κουβεντιάζουμε και τώρα άλλωστε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα θέματα να παραμένουν επίκαιρα, να μένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο πολιτικό πρόγραμμα. Αναφέρομαι στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μάλλον στη, χάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας. Έδωσε κάποιε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ερωτήματά μας, όμως είναι σημαντικό να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια, να δείξουμε ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τα μέλη της ενδιαφέρονται πάρα πολύ στο να υλοποιηθεί αυτή η χάρτα, να υπάρξει. Πρέπει να πούμε, να φανεί ότι οι Ευρωβουλευτές υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη συζήτηση. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μια συζήτηση στην Ολομέλεια πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα βάσει ερωτήσεων που θα υποβληθούν. Είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε τη δουλειά σε αυτόν τον τομέα και ταιριάζει και με την θέση της ίδιας της Επιτρόπου. Της δίδεται άλλη μια δυνατότητα να έρθει στο Κοινοβούλιο να εξηγήσει τις προθέσεις της και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Γι' αυτό υποστηρίζω το ερώτημα που προτάθηκε. Ευχαριστώ κύριε Φιγκορέδο. Και δίνω το λόγο στην κυρία Ισλέν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι πάντα πρέπει να τίθενται ερωτήματα. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συχνά, πολύ συχνά είναι ανεπαρκής και αόριστες. Δοθέντως όμως ότι τα ερωτήματα πάντα είναι χρήσιμα. Θα πρέπει να πούμε ότι αν θέσουμε αυτά τα ερωτήματα θα υπογραμμίσουμε και τη σημασία που έχει αυτό το θέμα για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Αυτό το έγγραφο της Επιτροπής είναι ανακοίνωση. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και έχει σαν υπότιτλο «Χάρτα των γυναικών» ή «Χάρτα χάρτης για τι Γυναίκε. Δεν έχω το κείμενο στα γαλλικά. Θα έπρεπε να συμπληρωθεί να είναι η χάρτα και δικαιώματα της γυναίκας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε μια χάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας, διότι έχουμε μια χάρτα δικαιωμάτων του ανθρώπου, των ανθρωπίνων όντων. Και μέχρι νεοτέρας οι γυναίκες παραμένουν ανθρώπινα όντα δεν θέλουμε μια χάρτα δικαιωμάτων της γυναίκας. Επειδή πρότεινε κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανε μια ανακοίνωση απλώς με αυτόν τον υπότιτλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάπως α, α, αξιοπρεπή που έχει κύρος. Πρέπει να επιπλώσει, να στολίσει την πρότασή της. Και πρότεινε να την εξοπλίσει αργότερα. Να υποβληθεί προφορική ερώτηση τώρα επ' αυτού του εγγράφου που έχει κάποιες σελίδες είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την ούτως αποκαλούμενη χάρτα. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα. Θα είναι αντιπαραγωγικό και να μην μιλάμε για χάρτα δικαιωμάτων της γυναίκας. Διότι δεν το πρότεινε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου στις εκθέσεις που ψηφίσαμε, αυτές τις εκθέσεις τις ατέρμονες που είναι ακατανόητες και κανείς θα τη διαβάσει, και αναφέρεται και εκεί μια χάρτα ε, δικαιωμάτων της γυναίκας. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν είναι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Έχουμε χάρτα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στα, έχει την έννοια του άντρα, έχει του, του, ε, του υπονοεί ανδρικό φύλλο, ενώ είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Λοιπόν, και δεκάδες χρόνια χρειάστηκαν, αυτοί που έχουν ηλικία μου το ξέρουν, για να έχουμε τα ανθρώπινα, ε, να έχουν ίσα δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα ο άντρας και η γυναίκα. Και θέλετε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για τα δικαιώματα της γυναίκα, κάτι που δεν πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το εγχείρημα, διότι θα κάνουμε ό,τι χειρότερο ε, είναι αντιπαραγωγικό όσον αφορά την ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Για τις απόψεις αυτές και δίνω το λόγο στην κυρία Γιάννα Κουδάκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μερικές φορές δεν μ' αρέσει να είμαι στην Επιτροπή αυτή, αλλά είμαι ακόμα εδώ και αγωνίζομαι. Κυρίες μου, αν σας δώσω ένα κουτί με σοκολάτες, το ανοίγετε και λέτε, πριν δείτε καν τι έχει μέσα, θα πείτε ότι α, δεν το θέλω αυτό. Και λέτε στον άνθρωπο που σας δίνει το δώρο τι θέλετε να περιέχει το κουτί. Η Επίτροπος ήρθε και μας είπε τι θα κάνει και πότε θα υποβάλει απάντηση. Γιατί βιαζόμαστε λοιπόν, γιατί τις πρόχνουμε. Γιατί προσπαθούμε να δείξουμε την ε, δύναμή μας. Διότι σας ε, ε, διαβεβαιώ, όταν προσπαθεί να δείξει κανείς τη δύναμή του, είναι επειδή δεν έχει μυς. Πιστέψτε με, εάν σπρώξουμε την ε, Επίτροπο, εάν την πιέσουμε, ε, δεν θα ε, συνεργαστεί πολύ καλά και δεν την κατηγορώ κιόλα. Α περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι απαντήσει τη όταν θα είναι έτοιμη και να προχωρήσουμε από εκεί. Αλλά το να ψηφίσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να στείλουμε προφορική ερώτηση, πιστεύω ότι θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για τι εργασίε μα. Εγώ προτείνω να αφήσουμε την ερώτηση για κάποια άλλη φορά. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει καλύτερα. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας. Να συνοψίσουμε. Υπάρχει διάσταση απόψεων Ίσως όχι όσον αφορά το στόχο, αλλά όσον αφορά και όχι για τη γνωμοδότηση για ε, τον ε, χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για το πώς ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. Από τη συζήτηση κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για υιοθέτηση προφορικής ερώτησης. Άκουσα τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ μια προφορική ερώτηση. Γι' αυτό προτείνω έναν πιθανό συμβιβασμό να εξετάσουμε τη δυνατότητα υποβολής τροπολογίας για την έκθεση της κυρίας Φιγερέιδο όταν συζητηθεί στην Ολομέλεια. να προτείνουμε κάποιο κείμενο για τους συντονιστές. Δεν θα το αποφασίσουμε αυτό σήμερα, διότι από ό,τι κατάλαβα ε, δεν ε, υπάρχει πλειοψηφία υπέρ λήψης απόφασης σήμερα. Υπάρχει κανείς που έχει παρατήρηση για την πρότασή μου να μην ψηφίσουμε σήμερα σχετικά με προφορική ερώτηση. Κυρία Κορνέλησεν, παρακαλώ. Συμφωνώ να μην ψηφίσουμε σήμερα για την προφορική ερώτηση. Δεν ξέρω ποια, η, τι, ποια είναι η πλειοψηφία, διότι η ΑΕΛΤΕ λείπει ολοκληρωτικά και συνήθως ε, αυτοί ε, κρατάνε την αποφασιστική ψήφο στα χέρια τους. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών. Είναι καλό που ακούσαμε τις απόψεις άλλων στην Επιτροπή μας και ίσως μπορέσουμε ως συντονιστές ε, το απόγευμα να εξετάσουμε διαφορετικές λύσεις, διάφορες λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλησεν. Κύριε Ιουβάν, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ακούσαμε τις απόψεις τις διάφορες και νομίζω ότι καλύτερα να ψηφίσουμε τώρα για να ακούσουμε την άποψη της ε, Επιτροπής μας τώρα. Υπέρ κατά. E, pani Przewodnicząca, uważam, że nie ma obowiązku przeprowadzania głosowań. No jeżeli... Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε. Άμα θέλουμε να το συζητήσουμε κι άλλο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε σήμερα. Mrs. Κυρία Λούλινγκ. Και εγώ λέω να ψηφίσουμε. Αρκετά μέλη ζήτησαν ε, να λάβουμε να ψηφίσουμε. Το θέμα υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει επιθυμία για ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σχετικά με την προφορική ερώτηση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι, η ερώτηση, ότι το θέμα υπάρχει στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών για σήμερα το απόγευμα. Είμαι πεπισμένη ότι θα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που θα πρέπει να συζητηθούν και ότι το θέμα θα ε, ξανασυζητηθεί ε, στην Επιτροπή μας. Αλλά θα ψηφίσουμε. Η κυρία Σβένσκι, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς είμαστε αρκετοί για να ψηφίσουμε. Ναι, έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Είμαστε έτοιμες να ψηφίσουμε με ανάταση χειρός. Όσοι θέλουν να εγκρίνουμε προφορική ερώτηση, παρακαλώ ψηφίστε τώρα. ποιοι απορρίπτουν προφορική ερώτηση. Παρακαλώ. Υπάρχει πλειοψηφία που απορρίπτει την υποβολή προφορικής ερώτησης. Μπορούμε πάντα να ε, υποβάλουμε προφορική ερώτηση στο όνομα κάποιου συνασπισμού. Προχωράμε στο θέμα 14 της ημερήσιας διάταξης. Punkten 14 Σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Ε, ο ρόλος του ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της στόχιας και για την πρόθεση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμού στην Ευρώπη. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρίαση. Θα έχουμε συζήτηση με αφορμή την έκθεση της κυρίας Φιγερέιδο ε, προς την Επιτροπή Απασχόλησης για το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος. Καλέσαμε την κυρία Φιγερέιδο για να μας εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα. Δίνω το λόγο στην κυρία Φιγερέιδο. Παρακαλώ και παρακαλώ και ταυτόχρονα παρακαλώ τους βουλευτές που εγκαταλείπουν την αίθουσα, να μην ε, συζητάνε μεταξύ τους μέσα στην αίθουσα. Όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα, θέλουμε να ακούσουμε την κυρία Φιγεράιδο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν μακρύ το πρωινό και καταλαβαίνω που φεύγουν αρκετοί από την αίθουσα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέμα που συζητείται στην Επιτροπή Απασχόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το ευρωπαϊκό έτος της καταπολέμησης της φτώχειας. Και τα στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά τρομακτικά. Τα στοιχεία όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρόνια μετά την ανακοίνωση στρατηγικής της Λέγαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την εκρίζωση της ένδυας, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός αποκλεισμός και φτώχεια στην Ευρώπη. Στην έκθεσή μου, ε, στο τελευταίο τμήμα της, περιέχονται δύο πίνακες που πιστεύω μιλούν από μόνοι τους. Δείχνουν πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Αυτοί οι πίνακες συμπεριλαμβάνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Eurostat που δημοσιεύτηκαν ε, φέτος βλέπετε σαφώς από τα στατιστικά στοιχεία ότι η φτώχεια σε σχετικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τη γραμμή, το όριο της φτώχειας και το κίνδυνο της φτώχειας, αφορά περίπου το 17% του πληθυσμού. Περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Μπορούμε να πούμε ότι η φτώχεια πλήττει 85 εκατομμύρια ανθρώπους συνολικά. Αυτά τα στοιχεία αφορούν το Δεκέμβριο του 2008. Δεν υπάρχουν πιο επίκαιρα στοιχεία και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πέρσι ήταν ο πιο σημαντικός χρόνος, η πιο σημαντική χρονιά όσον αφορά την κρίση. Και τώρα περνάμε από τις σοβαρές συνέπειες αυτής της κρίσης που πλήττει τη ζωή των ανθρώπων, η ενεργία έχει επιδεινωθεί, η πρόσκαιρη απασχόληση αυξάνεται, η μισθή είναι χαμηλή αρκετές χώρες ε, εισάγουν μέτρα λιτότητας με περικοπές όσον αφορά τα συστήματα ε, πρόνοιας. Πιστεύω ότι αυτά τα αριθμητικά στοιχεία θα έχουν ε, επιδεινωθεί σημαντικά από όταν έχουν ληφθεί αυτά τα στοιχεία. Αλλά ήδη και αυτά τα στοιχεία που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι αρκετά άσχημα. Και κάποια τμήματα του πληθυσμού πλήττονται όλους ιδιαίτερως. Βεβαίως τα παιδιά και οι νέοι. 20% είναι ο μέσος όρος. Σε ηλικία από 0 έως 17, που είναι κάτω από τη γραμμή της φτώχειας. Όπως βλέπετε, σε κάποιες χώρες αυτό το στοιχείο φτάνει μέχρι το 33% στην Ρουμανία, 20% στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία, σε αρκετές χώρες. Οπότε η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική. Διότι τα παιδιά και οι νέοι εκτίθενται δυσανάλογα στη φτώχεια. Και αυτή είναι η κατάσταση μετά τις κοινωνικές μεταφορές. Εάν ήταν πριν, αν ήταν παλιότερα τα στοιχεία, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Βλέπετε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μεταφορές. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πάνω από 65, πάρα πολλές γυναίκες. Σίγουρα θα το είδατε αυτό από κάποιες μελέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη σελίδα 9 της εκθέσεώς μου βλέπετε κάποια στοιχεία. Εκεί αναφέρεται ότι για τους ηλικιωμένου, ακόμα και μετά τη μεταφορά των κοινωνικών δικαιωμάτων, πάνω από 20% είναι κάτω από, την, το όριο της φτώχειας ή κινδυνεύουν να περάσουν αυτό το όριο. Και αν δείτε πιο συγκεκριμένα τις γυναίκες, 27% του, των γυναικών είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Μετά 18% με τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα για τις γυναίκες. Αλλά για τις ηλικιωμένες γυναίκες τα πράγματα είναι χειρότερα. Υπάρχει και ένα νέο φαινόμενο που δεν υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας. Ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ακόμα και όταν εργάζονται και έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, 20% εκείνων που κινδυνεύουν να περάσουν τώρα όριο της είναι αυτοί που εργάζονται. Η δουλειά δεν απαραίτητα μια απάντηση κατά της φτώχειας. Βλέπετε σε κάποιες χώρες όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Πορτογαλία, ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. 12%, 14% ε, στην Ελλάδα, Ρουμανία 17% από τους εργαζομένους κινδυνεύουν να περάσουν τη γραμμή της φτώχειας ή μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι στη φτώχεια, στα όρια της φτώχειας. Χαμηλή μισθή, ε, προσωρινή απασχόληση, σε κάποιες χώρες δεν είναι λύση αυτή για την καταπολέμηση της ένδυας. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Παρέθεσα αυτά τα στοιχεία για να δείξω τη σημασία που έχει κρατική παρέμβαση και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα Αυτά τα τελικά στοιχεία που παρουσίασα είναι μετά τα κοινωνικά επιδόματα, αλλά εκπονήθηκε μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει αυτή η μελέτη ότι πριν αυτά τα κοινωνικά επιδόματα ο κίνδυνος της φτώχειας για τα άτομα κάτω από 18 ετών είναι 33%. Για πάνω από 65 ετών είναι 24%. 25% για τους άντρες και 27% για τις γυναίκες, μετά από τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα που χορηγούνται. παρέθεσα κάποιους μέσους όρους, αλλά τα επίπεδα είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτό που βρίσκεται στην έκθεση είναι ότι λάβαμε υπόψη τα αίτια της φτώχειας, τις διάφορες μορφές που λαμβάνει η φτώχεια. Αναφέραμε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει πολλαπλός κίνδυνος, πολλαπλής διάκρισης ούτως υπήν, μετανάστες, γυναίκες, γυναίκες μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες με αναπηρίες. Υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις και παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στο κίνδυνο. Αναφέρθηκα σε διάφορα, σε διάφορα τμήματα του πληθυσμού, η φτώχεια όμως είναι πολυδιάστατη δεν εξετάζεις μόνο το εισόδημα, πρέπει να δεις και ποια είναι η δυνατότητα πρόσβασης στις διάφορες υπηρεσίες. Δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. Όταν όμως ο κόσμος δεν έχει ε, χρήματα, δεν έχει πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες, χρειάζονται δημόσιες υπηρεσίες συνεπώ. οι κρατικές υπηρεσίε που επιτρέπουν στου ανθρώπου να έχουν καλό επίπεδο θέρμανση, παιδεία, υγεία κλπ. Υπάρχει ένας πίνακας του Eurostat για την στέρηση, για την έλλειψη διαφόρων υλικών αγαθών. Ε, έχω παραθέσει αυτά τα στοιχεία στον πίνακα 2 της εκθέσεώς μου, αυτά τα στοιχεία του Eurostat. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει τους αναγκαίους πόρους για να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του ή για να έχει ένα πλήρες γεύμα κάθε μέρα. Δεν έχει χρήματα να πληρώσει για μια εβδομάδα διακοπών, να φύγει από το σπίτι του. Δεν μπορεί να έχει γιοταχή. υπάρχουν ποσοστά που αναφέρονται για κάθε χώρα και αυτά τα ποσοστά είναι άκρως ανησυχητικά θα έλεγα. Νομίζω ότι θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο διαφορετικά ζητήματα. Θέρμανση και ένα πλήρες γεύμα την ημέρα. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Σε διάφορες χώρες, βλέπετε τα στοιχεία, πάνω από 30% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις δύο πολύ βασικές υπηρεσίες, που είναι ουσιοδέστατες υπηρεσίες για την ελάχιστη αξιοπρέπεια της διαβίωσης. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ στον κατάλογο των χωρών που έχουν αυτό το πρόβλημα, αλλά ο πίνακα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι επιτρέπει να δει κανεί ότι η φτώχεια έχει πτυχές που ξεπερνούν το απλό θέμα του εισοδήματος. δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν τρώει κανονικά ε, την κάθε μέρα υποφέρει από πείνα και ότι ίσως διατρέχει κίνδυνο ε, πείνας, ε, αλλά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν σε κάποιες χώρες υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν καν να φάνε ένα αξιοπρεπές γεύμα, ένα κανονικό γεύμα την ημέρα. Αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βέβαια, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην παιδεία, στην κατάρτιση, στα συστήματα απόδοσης δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα έπρεπε να εμπεριέχονται σε δημόσιες πολιτικές που ανταποκρίνονται στην πολυδιάστατη υφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι φτωχοί δεν αποκλείονται απαραίτητα. Υπάρχουν διάφορες στοιχές που πολύ συχνά συγκλίνουν αλλά πτυχές που διαφέρουν μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που δεν αποκλείονται, αλλά είναι πολύ φτωχοί γιατί είναι πολύ χαμηλόμιστοι. Ε, μπορεί να έχουν προσωρινή, να ανασταθεί οι συνθήκες εργασίας τους. Να μην έχουν μόνιμη εργασία. Πρέπει να διαφοροποιούμε με προσοχή όμως τα διάφορα αυτά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το πλαίσιο όσον αφορά τις αμοιβέ, τους μισθούς και την αξιοπρεπή εργασία. Και βέβαια οι γυναίκες επηρεάζονται όλο ιδιαίτερω από όλα αυτά που ανέφερα. Πρόσβαση στη στέγαση. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πρόσβαση στι συντάξει. Συντάξει που να επιτρέπουν στον κόσμο να ζει με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που ε, πλήττει τις γυναίκες με χαμηλό μισθό, διότι πλήττονται διπλά. Και από τα θέματα τα συνταξιδοτικά και από το πρόβλημα της γύρανσης. Υπάρχουν τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε μισθό ούτε σε σύνταξη. Οι μισθοί και οι συντάξει είναι τόσο χαμηλά που δεν μπορεί να ζήσει κανεί αξιοπρεπώ. Για αυτού του ανθρώπου λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα. Βέβαια, ελάχιστο εισόδημα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα που εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Πρέπει να συνοδεύουμε το ελάχιστο εισόδημα με άλλες πολιτικές οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων που, δίνει, που θα δίνουν αυτοί οι τομείς, θα δίδεται πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορούν να απολαμβάνουν τα βασικά του ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το περίπλοκο θέμα του ελάχιστου εισοδήματο. Θα μπορούσαμε να θέσουμε κατοποκοπήν ε, ελάχιστο εισόδημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήταν καλή ιδέα. Το ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάθε χώρα ελάχιστο ημερομίσθιο σε εθνικό επίπεδο, ελάχιστο επίπεδο τιμών ε, στη χώρα, πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Όμως, όμως θα μπορούσαμε να έχουμε ισχυρότερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό από αυτόν που έχουμε τώρα. Το 1997 αναφέρθηκε η ανάγκη για ένα ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα και αυτή η συζήτηση λαμβάνει η χώρα τώρα στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει, πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή πολιτικών στήριξης για ελάχιστα εισοδήματα σε χώρες όπου αυτό θεωρείται ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε μια πολιτική συνοχή που φάνηκε ότι ήταν ανεπαρκέστατη όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που συζητούμε σήμερα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και ποιοι θα είναι οι μακροοικονομικοί προσανατολισμοί για να ανταποκριθούμε στην όλη κατάσταση. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φιγουρέιντο πολύ διεξοδική η παρουσίαση της έκθεσής σας. Αγωνίζεστε πάρα πολύ για την καταπολέμηση της φτώχειας και κυρίως ε, της φτώχειας των γυναικών. Υπάρχει κανείς που θέλει να κάνει σχόλιο? Αν όχι, έχουμε φτάσει στο 15. Τη σημερινή ημερήσια διάταξη που είναι τα διάφορα. Α, κυρία Κώστα. Πολύ σύντομα, διότι έχει περάσει η ώρα και έχουμε μείνει λίγοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Φιγκουερέιδο για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και τη σημαντική έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων, ε, ε, μα διαπαρακολουθήσουμε τι εργασίε τη Επιτροπή Απασχόληση, στην οποία είμαι αναπληρωματικό μέλο. Είναι καλό και σκόπιμο να θεωρείτε, να εξετάζετε το θέμα στην Επιτροπή Γυναικών, διότι γνωρίζουμε πως το πρόσωπο της φτώχειας και στον κόσμο και στην Ευρώπη έχει, είναι γυναικείο πρόσωπο. Να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Είναι σαφές, σαν υπόθεση, ότι είναι πολυδιάστατη φτώχεια, είναι πολλοί παράγοντες και είναι πολύ χρήσιμο, όπως λέει στο σημείο 7 και 8 της εκθέσεως, ότι πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό το έτος το ευρωπαϊκό, να βρούμε ε, συγκρίσιμους δείκτες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τους δείκτες φτώχειας, απόλυτης σχετικής φτώχειας και να δούμε και ποιοι άλλοι παράγοντες που να λαμβάνονται υπόψη. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι το ελάχιστο εισόδημα είναι κάτι που πειραμιστήκαν πολλές χώρες με αυτό και η χώρα μου η Ιταλία για κάποια χρόνια πειραματίστηκε με αυτό. Δυστυχώς δυσμονήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση ελάχιστο εισόδημα ένταξη. Κάποιε περιοχέ και κάποιε πόλει πειραματίστηκαν και θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε σύγκριση μελετών που έγινε σε διάφορε χώρε. Πώ λειτουργήσε θετικά, αρνητικά αυτό το μέτρο. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να, να δούμε δύο πτυχέ. Πρώτα απ' όλα, το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να είναι συμπληρωματικό, όπω είπε η κυρία Φιγκερέιδο. Να συμπληρώνει άλλα μέτρα ήταν πάντα μια ανησυχία ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να μειώσει τη διαθεσιμότητα για να δεχτεί κανείς προτάσεις κατάρτισης ή εργασίας. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε και πακέτα εντός εισαγωγικών για επίτευξη στόχων. Μείγμα ελαχίστου εισοδήματος, δυνατότητας κατάρτισης, προσανατολισμού και δυνατότητας πρόσβασης στην εργασία. Θα πρέπει να βρούμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση και διατύπωση. Δεύτερον, κάτι που συνδέεται πάρα πολύ με την ένταξη είναι με το, άτομο, το ξεχωριστό άτομο. Κάποιοι συνάδελφοι το είπαν αυτό και εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τα παιδιά και τη φτώχεια των παιδιών και των ανηλίκων θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το οικογενειακό εισόδημα. Που είναι ένα οικογενειακό εισόδημα όταν μια οικογένεια έχει μόνο ένα εργαζόμενο, μόνο ένα εισόδημα ή αν είναι μονογονική οικογένεια και αυτό σε σύγκριση με ε, ε, οικογένειες που έχουν πολλαπλά εισοδήματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα οικογενειακά εισοδήματα. Νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που θα να ακολουθήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό που λέω όσον αφορά αυτό το θέμα που θα μπορούσε να τιμήσει το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και να είναι και ευκαιρία να γίνουν μεγάλε διαβουλεύσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των διαφόρων ενώσεων και συνδέσμων που ασχολούνται με αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο, ζητώντα από τα κράτη-μέλη και από του βουλευτέ ενδεχομένω να βοηθήσουμε τόσο ώστε να γίνει μια διερεύνηση τι γίνεται ή να υποβληθούν κάποιε προτάσει από πλευρά μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η διαβούλευση αυτό το χρόνο και θα ήταν ενδιαφέρον εάν πάνω σε αυτό το θέμα ζητήσουμε πολύ περισσότερες δεσμεύσεις, πιο επίσημες δεσμεύσεις, ίσως και μια οδηγία πάνω σε αυτό, διότι πιστεύω ότι αξίζει μια πρωτοβουλία που θα οδηγήσει τα κράτη-μέλη να εθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα, διότι η φτώχεια, η αύξηση των ανισοτήτων, ε, είναι κάτι, αυτές οι τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές δεν είναι κάτι που, την, ε, που τιμά την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Κώστα για τις απόψεις σας αυτές. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει στις 24 Ιουνίου και να ευχαριστήσω και πάλι την υπεύθυνη για την Επιτροπή Απασχόλησης για το θέμα της καταπολέμησης της στόχιας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε... Α, η κυρία Φιγερέιδο θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα για τα σχόλιά της. Στο σχέδιο έκθεσης τονίζουμε ιδιαίτερα όσους ζουν στη φτώχεια και τους οργα... τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν. και βλέπουμε σε ποιου τομεί μπορούν να συμμετέχουν αυτοί, αυτές οι οργανώσεις. Πριν από 10 χρόνια εγκρίναμε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και εγώ ήμουν συγγήτρια τότε και μία από τις προτάσεις που είχα κάνει και έγινε αποδεκτή είναι μία ετήσια συζήτηση με όλους τους, ε, όλες τις οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις ε, και άλλες για την καταπολέμηση της φτώχειας και αυτό γίνεται. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές που δεν λειτουργήσαν τόσο καλά, άλλες πτυχές του προγράμματος αυτού. Και εξού και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Κάποιες από τις τροποποιήσεις που εγώ ίδια θα υποβάλω, θα λαμβάνουν υπόψη κάποιες από τις προτάσεις που εγκρίθηκαν πριν από 10 χρόνια τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να είναι πιο επιτυχές και να, και, να είναι πιο επιτυχής και η ετήσια συζήτηση που έχουμε για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και άλλα προγράμματα. Αλλά βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει και εκείνη περισσότερα. Πρέπει να λάβουμε περισσότερα στοιχεία. Οι μελέτες, ε, οι πιο πρόσφατες, ε, δεν καλύπτουν ε, την κρίση του τελευταίου έτους. Χρειαζόμαστε πιο πρόσφατα δεδομένα. Τον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή, μαζί με την Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της φτώχειας που είναι 17 Οκτωβρίου. Θέλουμε λοιπόν πιο πρόσφατα στοιχεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο πριν. Αυτό εμείς ζητούμε από πλευράς Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε την παρουσίασή μου, γιατί οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τη φτώχεια, πιο πολύ από τους υπόλοιπους και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα μέτρα που θα λάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγουρέιδο. Φτάσαμε στο τέλος διήμερης σκληρή δουλειά στην Επιτροπή μας. Η επόμενη μας συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου. Στο όνομα της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους, τους υπαλλήλους για τα πολύ καλά προετοιμασμένα έγγραφα για τη συνεδρίαση αυτή. Η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά και τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίω τη λήξη της συνεδρίασης.